Dear colleagues, I would like to start the meeting. Uh, uh, good morning everybody and uh, the first point on... Καλημέρα σας. Πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης ε, είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Δεν υπάρχουν προτάσεις για την τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης, γι' αυτό προτείνω να την εγκρίνουμε ως έχει. Δεύτερο σημείο, έγκριση των πρακτικών τη 27 η και 28 η Φεβρουαρίου και 19 η ε, και 20 η Μαρτίου του τρέχοντος έτους. Ω συνήθω έχουν μοιραστεί τα πρακτικά, οπότε ε, θα θεωρηθούν ως συγκεκριμένα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, εκτός και αν φυσικά υποβληθούν παρατηρήσεις και ενστάσεις. Άλλο σημείο το τρίτο, ανακοινώσεις της Προέδρου. Μία ανακοινώση έχω μόνο σε ό,τι αφορά την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης προκειμένου να παρασχεθεί αρρωγή στη Λιγουρία και τη Δοσκάνη μετά τις πλημμύρες του Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών εξετάζει το θέμα αυτό της ενεργοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης. Έχετε λάβει την πρόταση και ως συνήθως το ζήτημα είναι επίγον. Θα πρέπει να δώσουμε γνωμοδότηση. Τις τελευταίες τρεις ή τέσσερις φορές που ενεργοποίησαμε το Ταμείο Αλληλεγγύης, συνήθως ε, αναθέταμε στην Πρόεδρο την ε, αποστολή να στείλει επιστολή στην Επιτροπή Προπολογισμών λέγοντας ότι δεν έχουμε αντίρρηση με την ενεργοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύη. Αν συμφωνείτε και ε, αυτή τη φορά μπορώ να στείλω επιστολή προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών εκφράζοντας τη συμφωνία μας με την ενεργοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης. Δεν βλέπω να διαμαρτύρεται κανένας, οπότε μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης που προβλέπει συνέχιση της συζήτησης ε, για το γενικό κανονισμό. Θα εξετάσουμε το σχέδιο έκθεσης σε ό,τι αφορά τις κοινέ διατάξεις για τα ευρωπαϊκά ταμεία και την κατάργηση του κανονισμού 1083 του 2006. Πριν όμως δώσω το λόγο στους δύο συνεισηγητές, θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα αποτελέσματα της ε, συνεδρίασης της ομάδας εργασίας που έγινε χθες και που εξετάσαμε δύο θέματα, το χρονοδιάγραμμα για το πακέτο του Γενικού Κανονισμού και το συνολικό πακέτο και το κοινό στρατηγικό πλαίσιο. Συμφωνήσαμε λοιπόν στην ομάδα εργασία και αυτό σας προτείνω και εδώ να εγκρίνουμε να υποβληθεί η τελική έκθεση για το γενικό κανονισμό και να τη συζητήσουμε στις 29 Μαΐου εδώ. Οπότε προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών θα ξεκινήσει στη, να τρέχει στις 8 Μαΐου μέχρι 31η Μαΐου. Στόχος μας είναι να ψηφίσουμε, να γίνει μια ενδεικτική ψηφοφορία στην Επιτροπή μας στις 11 Ιουλίου, προκειμένου να θέσουμε εντολή στους συνεισηγητές για να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους εκπροσώπους του Συμβουλίου, προκειμένου η τελική ψηφοφορία να γίνει το φθινόπωρο. Δεν μπορώ να προβλέψω αν θα γίνει το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, πάντως η τελική ψηφοφορία θα γίνει το φθινόπωρο του 2012. Και μετά την τελική αυτή ψηφοφορία στην Επιτροπή μας, το φθινόπωρο, θα παραπέμψουμε την έκθεση αυτή στην Ολομέλεια. Συζητήσαμε και το σύνολο του πακέτου. Είπαμε να αντιμετωπίσουμε ως ενίο πακέτο όλες τις εκθέσεις και όλους τους κανονισμούς. Θέλουμε αυτή την συνολική προσέγγιση, να μην κατακαιρματίσουμε τη συζήτηση. Βέβαια, αν υπάρχει εύλογος λόγος ή έντονη επιθυμία κάποιου εισηγητή για συγκεκριμένο κανονισμό, φυσικά μπορούμε να είμαστε κάπως πιο ελαστικοί. Πάντως, γενικώ προτιμώ να εμείνουμε στην συνολική προσέγγιση, να την ε, χειριστούμε ως πακέτο. Τώρα, για το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, οι εισηγητές ε, θα μας υποδείξουν την ακολουθητέα διαδικασία. Δύο φορές το συζητήσαμε στην ομάδα εργασίας. Πάντως, οι εισηγητές πρότειναν και τα μέλη της ομάδας εργασίας συμφώνησαν το κοινό στρατηγικό πλαίσιο να αποτελέσει παράρτημα του Γενικού Κανονισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα έγγραφο εργασία, δηλαδή ένα έγγραφο χωρί νομική μορφή. Ω προς το χρονοδιάγραμμα, κανονίσαμε μια πρωτόλια εκδοχή του κοινού στρατηγικού πλαισίου να υποβληθεί στην Επιτροπή εδώ στις 8 Μαΐου αλλά η πλήρης η διεξοδική συζήτηση να γίνει στις 29 Μαΐου. Επίσης, όλες οι τροπολογίες που θα καταθέσουν τα μέλη της Επιτροπής ε, ΡΕΓΙ δεν αφορούν ε, τις εκθέσεις των εισηγητών, αλλά την ίδια την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπότε, αυτό να το έχετε υπόψη τα έγγραφα της Επιτροπής έχουν μοιραστεί ήδη από τον Οκτώβριο. Είναι διαθέσιμα. Βέβαια, θα έχουμε διαβουλεύσει και με τους εισηγητές και φαντάζομαι ότι στις 8 Μαΐου θα λάβουμε τις κατευθυντήριες γραμμές ε, και τους προσανατολισμούς των εισηγητών για να διευκολυνθείτε και στην κατάθεση τροπολογιών. Η διορία για τις τροπολογίες ξεκινά στις 8 Μαΐου και λίγη στις 31 Μαΐου. Αυτά ως προς τις ανακοινώσεις και τις εργασίες του, της ομάδας εργασίας. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Ελίζαβετ Στάτερ. Η Ευχαριστώ κύριε, κυρία Πρόεδρε. Χθε πράγματι συζητήσαμε αλλά δεν λάβαμε τελική απόφαση και επειδή η διαδικασία όπως την προτείνατε απαιτεί απόφαση της Επιτροπής μας και πρέπει να τηρηθεί και ο κώδικας διοντολογίας για τις σχέσεις με, την, με το Συμβούλιο θα ήθελα να παρακαλέσω τη Γραμματεία να συντάξει ένα σημείωμα που να περιλαμβάνει και τα τέσσερα βασικά θέματα που περιλαμβάνει ο, κώδικα, ο κώδικας διοντολογίας. δεν, μπορούμε, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε αν δεν κάνουμε πρώτα τα απαραίτητα αυτά βήματα. Η πρόεδρος δεν έχει μικρόφωνο δυστυχώς. Θα ήθελα να πω ότι ομάδα εργασίας ε, το συζήτησε με τους συγκητές γιατί οι συγκεκριτές θα αποφασίσουν τι μορφή θα έχει η έκθεσή τους και η σχετική απόφαση ε, θα γίνει σήμερα από την Επιτροπή, εκτός και αν υπάρχουν αντιρρήσεις ή αν έχετε διαφωνίες ως προς την προσέγγιση. Και στις ε, προθεσμίες. Αλλιώς οι προθεσμίες θα πρέπει να γίνουν σεβαστές. Τα όσα εξηγήσατε δεν επαρκούν για να συμπληρωθεί, να ε, λάβει μορφή δηλαδή ο κώδικας διοντολογίας. Γι' αυτό και προτείνω η γραμματεία να συντάξει το σημείο που εξήγησα προηγουμένω, ώστε να μπορέσει να συμπληρωθεί, να πληρωθεί, να γεμίσει ο κώδικας. Αυτά που λέτε εσείς είναι έκθεση, δεν είναι σχέδιο αποφάσεως. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα κριτήρια για το πώς συντίθεται μια διαπραγματευτική επιτροπή και ποια είναι η διαδικασία. Και παρακαλώ να τηρηθεί η διαδικασία. Άλλωστε δεν είναι και επίγον, δεν υπάρχει πρόβλημα να αναβληθεί απόφαση για την επόμενη συνεδρίαση, την οποία απόφαση μπορούν να προπαρασκευάσουν οι συντονιστές. Παρακαλώ λοιπόν να γίνουν τα απαραίτητα προπαρασκευαστικά βήματα. Εάν δεν συμβεί αυτό, τότε θα εμείς, εμείς θα προβούμε στα κατάλληλα διαβήματα. Θα θέλατε να αναφερθείτε σε κάποιον συγκεκριμένο κανόνα. Κοιτάξτε, ο κώδικα διοντολογία λέει ότι συμμετέχουν στη διαπραγματευτική επιτροπή όλε οι πολιτικέ ομάδε. Δηλαδή εκλέγονται τα μέλη τη επιτροπή και αυτό πρέπει να γίνει. Πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία, πρέπει να υποβληθεί γραπτό στην επιτροπή μα και να ληφθεί από αυτού απόφαση. Παρακαλώ λοιπόν να συμβούν αυτά τα οποία αιτούμε. Κατανοώ ότι αναφέρεστε στο σύνολο των διαπραγματεύσεων, θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό και θα εξετάσουμε και το αίτημά σας. Όπως είπα στην αρχή, υπάρχει μία πρόταση η οποία προέρχεται από τους εισηγητές και συζητήθηκε χθε από όλους όσους πήραν μέρος στην συνάντηση της ομάδας εργασίας που είναι ανοιχτή φυσικά σε όλους τους εισηγητές και σε όλους τους συντονιστές παρουσίασα εγώ τις συστάσεις χθες που είχαν συμφωνηθεί στην ομάδα και δεν υπάρχει κάποια διαφωνία. Έχουμε συμφωνήσει και στο χρονοδιάγραμμα. Σχετικά τώρα με το θέμα που έθεσε η κυρία Σουέτα, θα το διευκρινίσει η γραμματεία και θα δοθεί απάντηση μέχρι την επόμενη συνάντηση. Να δούμε τι ακριβώς πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Και φυσικά θέλουμε να γίνει σεβαστός ο κώδικας συμπεριφοράς. Καλώς, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις από ό,τι βλέπω. Μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 4. Δίνω το λόγο στους εισηγητές, δεν ξέρω πώς ακριβώς θα μοιράσετε τον χρόνο σας. Θα ομιλήσω την Αγγλική, λέει ο κύριος Βανίστελ γιατί και το αρχικό κείμενο ήταν στα Αγγλικά. Ξεκινώντας, θα ήθελα να πω σε όλους τους φίλους της Επιτροπής μας εδώ, γιατί εδώ είναι μόνο φίλοι της Επιτροπής, ότι το συγκεκριμένο θέμα γύρω από τους νέους κανονισμούς και το, δύο, το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο υπάρχουν τέτοιου είδους υποστήρικτες όπως υπάρχουν και υποστήρικτες της Προεδρίας, όπως υπάρχουν και υποστήρικτες της Επιτροπής και πάει λέγοντας. Λοιπόν, εμείς έχουμε πολύ συγκεκριμένες ευθύνες και μάλιστα θα έλεγα έχουμε ηγετική θέση και θα πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε όπως το κάναμε μέχρι τώρα. Θα πρέπει δηλαδή ε, με συγκεκριμένο τρόπο να ενημερώνουμε τους συναδέλφους μας οι οποίοι δεν ασχολούνται ειδικά με το θέμα και όλες τις άλλες επιτροπές που ασχολούνται λιγότερο με το θέμα. Πρέπει να είμαστε λοιπόν δραστήριοι, πρέπει να είμαστε διαφανείς και ήδη πριν από το καλοκαίρι να έχουμε ξεκαθαρίσει το πού βρισκόμαστε, το ποια είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή τη συγκεκριμένη σημαντική συζήτηση. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να συζητήσουμε σοβαρά με το Συμβούλιο, γιατί ξέρετε ότι η Προεδρία έχει έλθει και μας έχει πει ακριβώς τι πρόοδος έχει υπάρξει στο Συμβούλιο γύρω από αυτό. Μερικές φορές αντίθετα εμείς δεν είμαστε απόλυτα βέβαιοι για το τι είδους πρόοδο θέλουμε να κάνουμε. Και μερικές φορές δεν έχουμε εμβαθύνει όσο θα έπρεπε να εμβαθύνουμε. Είναι η τέταρτη φορά που συζητάμε λοιπόν το θέμα στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας έτσι ώστε να καταλήξουμε κάπου πριν από τις διακοπές. Έχουμε το κείμενο εργασίας, δέκα σημεία, το έχουμε συζητήσει σε βάθος και αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε σήμερα είναι να παρουσιάσουμε την πρώτη τροπολογία η οποία να συμβαδίζει θα έλεγα με τις δικές σας απόψεις και την αίσθηση που έχετε για τις συζητήσεις στις τελευταίες συναντήσεις μας. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε, ας ε, ε, συλλέξουμε τις απόψεις τις οποίες έχετε και ας τις μεταφράσουμε τις απόψεις αυτές σε ουσία μέσω της τροπολογίας. Να επαναλάβω αυτά τα οποία έχουν υποθεί για, την, για τον χρονισμό αν θέλετε. Υπάρχουν ε, ήδη κάποιες τροπολογίες σε αυτή τη φάση ουσιαστικά Εμείς θα προσπαθήσουμε να διευκρινίσουμε και να ενσωματώσουμε τις παρατηρήσεις σας. Σε μια δεύτερη φάση θα έχουμε συλλέξει όλες τις τροπολογίες μπροστά μας, θα έχουν μεταφραστεί οι τροπολογίες αυτές. Είναι στο τέλος, θα εξαντλήσουμε την περίοδο αυτή δηλαδή ε, έχει σημασία το κείμενο να μην μείνει μόνο στα αγγλικά, να έχει μεταφραστεί έτσι ώστε όλοι να μπορέσετε να λάβετε σοβαρά υπόψη το κείμενο. και να μπορέσετε έτσι να διαπιστώσετε το γιατί και το πώς εμείς έχουμε καταλήξει σε αυτές τις τροπολογίες. Δεν θα πρέπει, θα πρέπει μάλλον να αποφύγουμε να υπάρχουν επαναλήψεις να υπάρχουν περισσότερες τροπολογίες από όσες χρειάζονται και δεν πρόκειται για ουσιαστική εμπλούτιση της διαδικασίας αν κατατεθούν εκατοντάδες τροπολογίες βέβαια. Λοιπόν, ελπίζω να καταλήξουμε στην πρώτη ψηφοφορία τον μήνα Ιούλιο. Και μετά θα δούμε πώς θα συνεχιστεί η διαπραγμάτευση έχοντας κατά κάποιο τρόπο ελέγξει πλέον τις απόψεις μας. Αυτή είναι λοιπόν η άποψή μου. Κάποιες παρατηρήσεις τώρα. Αυτό που έχει σημασία είναι η συνοχή του κοινού αυτού στρατηγικού πλαισίου. Ήμουν στην Επιτροπή Ήτρε τη Δευτέρα και άκουσα ότι το κοινό αυτό στρατηγικό πλαίσιο δεν θα πρέπει να είναι τμήμα μιας κατεξουσιοδότηση πράξεως. Αντίθετα θα πρέπει να είναι κομμάτι μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας. Και τώρα έχουμε τις τροπολογίες που μας επιτρέπουν να το ισχυριστούμε αυτό. Υπάρχει λοιπόν τροπολογία η οποία αναφέρεται στις θέσεις τις οποίες περιλαμβάνει το κοινό στρατηγικό πλαίσιο στον τίτλο ήδη και σαν παράρτημα και στο κύριο κείμενο εμείς λέμε ότι το, η πρόταση αυτή, το κείμενο το οποίο εν πάση περιπτώσει εδώ προτείνεται, κατατίθεται, ε, είναι κάτι το οποίο θα αντικαταστήσει τον λεγόμενο κοινό κανονισμό. Αυτό έχει σημασία. Έχει σημασία για να δείξουμε ε, ποια είναι η νομοθετική ρύθμιση την οποία θέλουμε να βελτιώσουμε και να αντικαταστήσουμε. Πρόκειται για μια τροπολογία η οποία θα είναι οριζόντια θα έλεγα. Το συζητήσαμε αυτό στο έγγραφο εργασίας. Είπαμε ότι θα έχουμε και ένα νέο κείμενο στο άρθρο 2 το οποίο θα διευκρινίζει ακριβώς τη φύση αυτού του πλαισίου. Αυτό θα το κάνουμε με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε τουλάχιστον σε αυτή τη φάση να μπορέσουμε να εξηγήσουμε ήδη ότι καταθέτουμε ένα κείμενο σε αυτή τη φάση το οποίο σε επίπεδο νομικό δεν έχει φτάσει στο απαιτούμενο επίπεδο λεπτομέρειας. Ελπίζω όμως ε, στις 8 Μαΐου ήδη να είμαστε σε θέση να σας διευκρινίσουμε τα βασικά σημεία του περιεχομένου του κοινού στρατηγικού πλαισίου μέσω μιας διαδικασίας η οποία θα δίνει τη δυνατότητα να υπάρξουν αλλαγές, τροπολογήσεις κτλ. Να αναφερθώ τώρα στα άρθρα που έχουν σχέση με την αρχή της εταιρικότητας, το 4-4. Εμείς έχουμε ήδη ενισχύσει αρκετά την θέση των εκπροσώπων των περιφερειακών, τοπικών και δημοτικών αρχών σε σχέση με τους υπολείπους εταίρους και έχουμε ορίσει νομίζω καλύτερα τους όρους συμμετοχής των αρχών αυτών. Η σύμβαση η εταιρική, αναφέρομαι εδώ ιδιαίτερα στο άρθρο 13, είναι κάτι το οποίο διευκρινίζεται επιπλέον και προτείνουμε μάλιστα και μία τροπολογία η οποία να ενισχύει τις αρχές της εταιρικής αυτής σχέσης, να διευκρινίζει τα της προπαρασκευής και ε, σύνταξης της έκθεσης προόδου σε επίπεδο περιφερειακών στρατηγικών. Έχουμε επίσης καταθέσει ε, μια τροπολογία η οποία διευκρινίζει τις, ε, τη φύση των δραστηριοτήτων συνεργασίας και σε περιφέρειες υπηρετικές και σε περιφέρειες θαλάσσιες. Αυτά είναι κάποια επιμέρους σημεία τα οποία θα ήθελα εκ των προτέρων να διευκρινίσω και θα ήταν μάλλον θετικό σε αυτή τη φάση ήδη να ακούσουμε τις απόψεις κάποιων συναδέλφων σε μια πρώτη φάση που ασχολούνται με τέτοια συγκεκριμένα θέματα. Θα ήθελες ίσως να αναφερθείς τώρα σε κάποια άλλα σημεία τα οποία ίσως δεν αναφέρθηκα. Θέλει να κρατήσει κάποια μυστικά. Η Κώσταντς θέλει κάτι να προσθέσει. Όχι, όχι, μυστικά δεν υπάρχουν. Εμείς είμαστε τόσο διαφανείς και άλλωστε είναι σημαντικό για ένα τέτοιο εγχείρημα ένα τέτοιο δηλαδή πακέτο για την πολιτική συνοχή για τα επόμενα 7 χρόνια. Είναι τόσο σημαντικό αυτό. Άλλωστε όπως έχουμε διαπιστώσει και από παρελθούσες συζητήσεις, αυτές στράφηκαν πάντα όχι μόνο γύρω από την πολιτική συνοχή, αλλά και γύρω από την επίτευξη των στόχων Ευρώπης 2020, δηλαδή και στόχοι για το κλίμα και για τις απότατες περιφέρειες και για τα δημογραφικά. Είναι λοιπόν τόσο μεγάλη η δέσμη αυτή που ξεφεύγει και από τα όρια του απλού νομοθετικού κειμένου. Νομίζω ότι η φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ικανότητα ολοκλήρωσής της θα εξαρτηθεί από αυτές τις συζητήσεις. Και έχει δίκιο ο Λάμπερτ όταν λέει ότι χρειαζόμαστε και τους φίλους, τους φίλους της Προεδρίας και τους φίλους της ε, Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και θα τους χρειαστούμε όλους αυτούς τους επόμενους μήνες. Είναι απαραίτητο να ενταχθούν όλες αυτές οι συνεργασίες μέσα σε αυτή τη διάφανη, όπως είπα, διαδικασία. Μία συμπλήρωση για το κοινό στρατηγικό πλαίσιο. Συζητήσαμε βέβαια εάν όντως είναι το σκοπιμότερο να το βάλουμε σε ένα παράρτημα ή αν ίσως είναι καλύτερα να ζητήσουμε άλλο κανονισμό. Όμως, εάν το συνδέσουμε, εμείς θεωρούμε ότι αυτός ο γενικός κανονισμός θα αποτελεί την στέγη που θα καλύψει πέντε διαφορετικά ταμεία. Δεν μπορώ τώρα να βάλω πάνω από αυτή τη στέγη άλλη μία πιο μικρή, το strategic frame δηλαδή, που αυτό θα σημαίνει όμως εάν ζητήσουμε έξτρα κανονισμό για το CSF. Και γι' αυτό είπα να το βάλουμε στο παράρτημα. Η Κομισιόν νομίζω δεν έχει διάθεση να το κάνει. Γι' αυτό είπαμε εμείς θα καταθέσουμε πρόταση, θα καταθέσουμε τροπολογία για το CSF. Ασφαλώς ζητούμε πολλά από τους συναδέλφους, αλλά πολλές απαιτήσει έχουμε και από τους ίδιους τους εαυτούς μας. Διότι είναι πράγματι σημαντικότατη προσπάθεια να καταλήξουμε δηλαδή σε ένα έγγραφο μέχρι τον Ιούλιο όριμο για να ληφθεί απόφαση από αυτού σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά πρέπει να γίνει, διότι είναι κρίσιμος ο δρόμος αυτός για τα επόμενα 7 χρόνια της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω και ορισμένα άλλα θέματα για τα οποία έχουμε καταθέσει τροπολογίες και κυρίως τον τομέα της ελαστικότητας, η ευκαμψίας, επίσης οι τροπολογίες 61-66 που αναφέρονται στο άρθρο 87. Σε πολλές συζητήσεις τα είπαμε αυτά για πολυταμιακή, για πολυταμιακό μάλλον προγραμματισμό και χρηματοδότηση κλπ. Εάν επιτύχουμε να ψηφιστούν αυτά, τότε θα δώσουμε στις περιφέρειες μια δυνατότητα να αποφασίσουν οι ίδιες αν θέλουν αυτή την πρόσβαση στα πολλαπλά ταμεία και να μπορούν έτσι να εφαρμόσουν τα προβλεπόμενα από την πολιτική συνοχή με τρόπο εύκαμπτο. Αυτά νομίζω ότι θα συζητηθούν και τους επόμενους μήνες. Ελπίζω δεν έχω την υποστήριξή σας. Οι εισηγητές μετά από τις πολλές συζητήσεις έχουν συμφωνήσει, άλλωστε έχουν δει ότι υπάρχει μεγάλη συμφωνία για το ότι δεν θέλουμε να αποδεχθούμε το αποθεματικό επίδοσης που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη μορφή που το προτείνει. Έχουμε την εντύπωση ότι η ιδέα δεν είναι άσχημη αυτήν αλλά η εφαρμογή μέσω αυτού του εργαλείου δεν είναι κατάλληλη. Γι' αυτό και θέλουμε να προτείνουμε ε, αντίστοιχα τη διαγραφή του αποθεματικού επίδοσης κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει και στα διάφορα άρθρα και στις ε, διάφορες παραγράφους και εδάφια με κατάλληλες τροπολογίες και νομίζω ότι δεν είναι μόνο ότι θέλουμε ένα ανταγωνισμό για καλύτερα έργα, καλύτερα σχέδια, καλύτερη διεξαγωγή της πολιτικής, αλλά θέλουμε επίσης να μην δημιουργηθούν ανυπέρβλητα γραφειοκρατικά εμπόδια. Γι' αυτό προτείνουμε να αφαιρεθεί αυτό από την πρόταση της Κομισιόν. Το ίδιο προτείνουμε την αναφορά στη μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Να διαγραφεί αυτή. Από τις πιο απλές τροπολογίες. Λέει διαγράψτε το άρθρο 21. Διαγραφή το άρθρο 21. Πιστεύουμε ότι αυτή η μακροοικονομική αιρεσιμότητα ασφαλώς και είναι σημαντική. Δεν υπάρχει θέμα ότι οι χώρες μέλη οφείλουν να εξηγαίνουν τους προπολογισμού τους. Δεν τίθεται θέμα αυτό. Αλλά πρέπει να φέρουν την ευθύνη οι περιφέρειες για τις καταχρήσεις που ενδεχομένως κάνουν οι κυβερνήσεις, οι κεντρικές κυβερνήσεις. Και όπως βλέπουμε, η πολιτική συνοχή είναι το μοναδικό εργαλείο που προσφέρει επενδύσεις και ανάπτυξη στις χώρες μέλη. Όταν λοιπόν πάμε σε χώρες μέλη οι οποίες ούτως ή άλλως αντιμετωπίζουν δυσχέρειες και τους αφαιρούμε το εργαλείο αυτό, αυτό νομίζουμε ότι είναι λάθος. Γι' αυτό προτείνουμε διαγραφή, χωρίς να σημαίνει ότι δεν μπορούν να συνεχιστούν υφιστάμενα εργαλεία, όπως για παράδειγμα το Ταμείο Συνοχής, που όμως δεν αποτελεί τμήμα του Γενικού Κανονισμού και γι' αυτό δεν εμφανίζεται εδώ. Εδώ στην Επιτροπή Περιφερειακής Αναπτύξεως έχουμε συζητήσει κατ' επανάληψη για την αιρεσιμότητα εκ των προτέρων, ex ante conditionality. Οι εισηγητές πιστεύουν ότι αυτή η ex ante conditionality έχει νόημα, μπορεί να έχει νόημα, εάν βέβαια έχει άμεση σχέση με την πολιτική συνοχή, εάν δηλαδή αφορά άμεσα την πολιτική συνοχή να υπάρχουν άμεσες διασυνδέσει ανάμεσα στους σχεδιασμούς που γίνονται σε μια χώρα μέλος, τα έργα δηλαδή που σχεδιάζονται στην βάση της πολιτικής συνοχής και σχετική νομοθεσία. Και γι' αυτό έχουμε κάνει ορισμένες προτάσεις που αναφέρονται κυρίως, εμφανίζονται κυρίως στις ε, τροπολογίες 35-38 και 54-56. Και εκεί πρέπει να κάνουμε την απαραίτητη επεξεργασία για να περιληφθούν στα παρατήματα. Τώρα τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Αυτά νομίζω είναι σημαντικό νέο μέρος για την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο που θα φανούν εκεί πολύ περισσότερο Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να δράσουμε αποτελεσματικά, πώς μπορούμε να δαπανίσουμε πιο αποτελεσματικά δηλαδή τα ευρωπαϊκά κονδύλια και στις περιφέρειες και νομίζω ότι με τις προτάσεις μας όντως προωθούμε την ιδέα να χρησιμοποιηθούν χρηματοδοτικά εργαλεία για να ξεφύγουμε από τις καθαρές επιδοτήσεις, να προχωρήσουμε λίγο στην κατεύθυνση των δανείων Επίσης τα χρήματα αυτά να μπορούν να ανανεώνονται, να είναι ανανεώσιμα κεφάλαια. Αυτό επίσης είναι σημαντικό. Άλλωστε εν μέρη τα λέει αυτά και όλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της. Αλλά χρειαζόμαστε πάλι ξεκάθαρους κανόνες που να συναποτελέσουν τμήμα του κανονισμού, να ενταχθούν στον κανονισμό για τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε και εμείς κάνει ορισμένες προτάσεις για να προλιάνουμε το έδαφος έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε και κάποιες παραλήψεις σε κάποιους ορισμούς της Κομισιόν. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε κάνει και τις κατάλληλες τροπολογίες. Εάν εξετάσετε το πρώτο σχέδιο του κειμένου θα δείτε ίσως ότι έχουμε συζητήσει και πολύ περισσότερα πράγματα στην Επιτροπή και ότι εκφράσαμε πολύ περισσότερες επιθυμίες. Ο Λάμπερτ σωστά είπε ότι πρόκειται για ένα πρώτο μέρος και για μια πρώτη φέτα εντός εισαγωγικών των τροπολογιών και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να σας υποβάλουμε όλες τις υπόλοιπες στις 8 Μαΐου. Αλλά θα σας επιστήσω την προσοχή στο εξής, ιδίως για την απλούστευση, κάτι το οποίο μας απασχολεί πολύ ως θέμα, σε ορισμένα σημεία δεσμευόμαστε ακόμη, διότι παραλλήλως με τις συζητήσεις που διεξάγονται στην δική μας Επιτροπή, το Κοινοβούλιο διαπραγματεύεται τον δημοσιονομικό κανονισμό και τίθεται θέμα, για παράδειγμα, για μια αρχή πιστοποίησης. Μπορούμε λοιπόν να προτείνουμε εμεί τροπολογίες, αλλά ενδεχομένως αυτές να καταστούν άνευ αντικειμένου. Αυτή τη στιγμή υπάρξει απόφαση η συμφωνία με το Συμβούλιο, δηλαδή μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Εξαρτώμεθα λοιπόν από αυτή τη μελλοντική απόφαση, ώστε ακόμη δεν μπορούμε να συντάξουμε τίποτα σχετικά. Ελπίζουμε ότι τον Ιούνιο το Κοινοβούλιο θα καταλήξει σε μια τελική απόφαση όπως είπα, σε συνεργασία με το Συμβούλιο και θα δούμε τότε πώς θα αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, θεωρούμε ότι τον Ιούλιο, 7ο μήνα δηλαδή, θα πρέπει να διεξαχθεί συζήτηση στην Επιτροπή Περιφερειακής Αναπτύξεως για να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε πάλι με την Κομισιόν, να βρούμε τρόπους, να βρούμε δρόμους, να προωθήσουμε τα δικά μας ενδιαφέροντα για τη μελλοντική πολιτική συνοχή. Εν τέλει, λίγα σχόλια προς την κατεύθυνση της Κομισιόν. Ασφαλώς η Κομισιόν τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες πια έχουν γίνει, μας έχει υποστηρίξει πολύ. Μας έχει δώσει πληροφορίες, εξηγήσει, έχει προχωρήσει συζητήσεις μαζί μας για να εξεύρουμε τον σωστό δρόμο που προσπαθούσαμε άλλωστε να βρούμε για τη μελλοντική πολιτική συνοχής και ασφαλώς η Κομισιόν σε κάποια σημεία, όπως για παράδειγμα στο CSF, αλλά και για την ε, ευκαμψία ε, και για το αποθεματικό επίδοσης και ούτω καθεξής, φαντάζομαι ότι θα έχει πλέον απαυδίσει και θα λέει, μα τι κάνει επιτέλους το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όμως, νομίζω ότι μπορεί να είναι πεπισμένη η Κομισιόν ότι εμείς κάνουμε ορθές και λογικές προτάσεις. Και ελπίζω πολύ η Κομισιόν να φανεί να, ε, διατεθειμένη να μας υποστηρίξει, διότι θα είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακολουθήσει τον ίδιο αυτό δρόμο μαζί μας. Και νομίζω ότι το αξίζουν οι περιφέρειες να ε, γίνει αυτή η προσπάθεια. Και ειδικά για την ευκαμψία λέει ότι αυτό θα είναι αντίθετο με την συγκέντρωση των πόρων. Εγώ νομίζω ότι το αντίθετο θα συμβεί, διότι πρώτα-πρώτα υπάρχει μόνο μία δυνατότητα να βοηθήσουν οι χώρες μέλη της περιφέρειας και δεύτερο είναι και προς το συμφέρον των ίδιων των περιφερειών να προσπαθήσουν να τηρήσουν τους στόχους της Ευρώπης 2020 για το κλίμα, για την καταπολέμηση της φτώχειας, της ανεργίας. Και νομίζω ότι εάν θέλουμε να προσφέρουμε κάποια ευκαμψία σε όλη αυτή την ποικιλία των περιφερειών, με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνει, ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί και η συγκέντρωση των πόρων. Και σε ό,τι αφορά την μακροοικονομική αιρεσιμότητα, αυτό βεβαίω πάσχει από το ότι οι μεν ε, πιστεύουν το ένα, οι άλλοι το άλλο. Υπάρχουν δύο διαφορετικέ θέσει. Όταν η ίδια η Κομισιόν λέει ότι δεν θέλουμε καν να χρησιμοποιήσουμε το μέσον αυτό, έχει μόνο αποτρεπτικό χαρακτήρα, τότε μπορεί κανεί να πει ότι μπορεί να προσφέρει και θετικά επιχείρηματα, να προσφέρει θετική υποστήριξη στι χώρε και όχι να κρεμά την δαμόκλειο σπάθη πάνω από τα κεφάλια του επίδραση άλλωστε προς τα έξω είναι και ψυχολογική. Αν δουν δηλαδή οι περιφέρειες ότι τις υποστηρίζουμε, ότι ανοίγει και μια πρόσβαση σε μια συζήτηση για το πώς θα αντιμετωπίσουμε δηλαδή με διαφορετικό τρόπο τις, δυσκολ... τις δημοσιονομικές δυσκολίες από το να τους πούμε αν δεν κάνεις αυτό τότε θα σου κάνω αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι ακόμα και για παιδαγωγικούς λόγους είναι πολύ απλούστερο να τους προσφέρουμε μια λογική πολιτική και χώρες οι οποίες είναι πραγματικά σε δυσκολίες να δουν ότι μπορούμε να τις βοηθήσουμε. Ελπίζω τις επόμενες εβδομάδες, την επόμενη εβδομάδα πρώτα-πρώτα, θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε και να προχωρήσουμε. Ελπίζω και αυτό το απευθύνω τώρα και στο Συμβούλιο. Ελπίζω το Συμβούλιο να μην προσπαθήσει, να μην συνεχίσει μάλλον να προσπαθεί να απαξιώνει την νομοθετική εργασία του Κοινοβουλίου βάζοντας όλα στο καλάθι των διαπραγματεύσεων για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και να πει ότι εμείς τώρα θα διαπραγματευτούμε για τον προπολογισμό, θα λάβετε αβγ στα τάδε σημεία και δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε παραπέρα για πράγματα τα οποία ωστόσο εντάσσονται στη συναπόφαση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν είναι αποδεκτό κάτι τέτοιο και γι' αυτό παρακαλώ προς το συμφέρον όλων και των περιφερειών να γίνει σαφής διάκριση ανάμεσα στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και στο νομοθετικό έργο, το οποίο προσεγγίζουμε από κοινού, όχι το Κοινοβούλιο κατά του Συμβουλίου, από κοινού. Και από κοινού προβλέπεται στην συνθήκη της Λισαβόνας. Η δημοκρατία σημαίνει εν τέλει ότι όλοι υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους και άλλωστε και προς τα έξω πρέπει να φανεί καθαρά ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα όργανο εκλεγμένο το οποίο νοιάζεται, φροντίζει τα ενδιαφέροντα και συμφέροντα των πολιτών και των κέντρων και της περιφέρειας. Δεν μπορούν να τα ρίξουν όλα μαζί σε ένα διαπραγματευτικό καλάθι το οποίο συζητείται και γίνεται αντικείμενο διαπραγμάτευσης open-end πίσω από κλειστές θύρες. Ελπίζω λοιπόν οι θέσεις αυτές του Κοινοβουλίου να γίνουν σεβαστές και να γίνει στη βάση αυτή η διαπραγμάτευση. Ευχαριστώ Κωνσταντζα. Θα ακούσουμε τους κέντες ηγητές τώρα, τώρα. Πρώτα ο κύριος Γκοτσμάνης. Ευχαριστώ. είμαι σε μηχανία γιατί δεν νομίζω ότι είμαστε σε οριστική φάση της διαδικασίας γιατί τελικά σε τροπολογίες θα καταλήξουμε μόνο. Πάντω θα ήθελα να συγχαρώ τους συγητές που πραγματικά επιτέλεσαν πολύ αξιόλογο έργο. Γιατί αν διαβάσουμε προσεκτικά τις τροπολογίες, βλέπουμε ότι λαμβάνουν υπόψη τη πλειοψηφία των σχολείων. Εγώ θα εκφράσω τη γνώμη μου για πέντε θέματα. Στην τροπολογία 2, όπου είπαν οι συνεισηγητές ότι κάτω χώρες δεν θα μπορούν ανεξάρτητα από τις περιφέρειες και την τοπική ε, αυτοδιοίκηση να κάνουν τις εταιρικές, να δημιουργήσουν εταιρικέ σχέσεις με βάση το κανονιστικό πλαίσιο κτλ. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη δηλαδή η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεύτερον, για το αποθεματικό επίδοσης. συμφωνώ με την κατάργηση αυτού του αποθεματικού. Γιατί αν επιτρέψουμε τη διατήρησή του, τότε εκείνες οι διοικήσεις που θα, μπορούν προσπαθήσουν, που θα είναι επιφορτισμένες με την εφαρμογή των προγραμμάτων, θα προτιμήσουν πιο απλά και λιγότερο περίπλοκα σχέδια. Οπότε θα αρχίσουν μεταφορές κονδυλίων από τα πιο περίπλοκα και βαριά προγράμματα και σχέδια στα πιο light, στα πιο ελαφρά, οπότε η προστιθέμενη αξία θα είναι λιγότερη. Η τροπολογία 7 κατά τη γνώμη είναι πιο σημαντική γιατί η αιρεσιμότητα που συνδέεται με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα ληφθεί υπόψη, αλλά σε συνδυασμό με την απορρόφηση από το Ταμείο Συνοχής κτλ. Συμφωνώ απόλυτα με την προσέγγιση αυτή, γιατί διαφορετικά θα μπορούσαμε τον κατονισμό αυτό να αντικαταστήσουμε αυτά που θα κυρώσουν τα κοινοβούλια μέχρι τα μέσα του έτους. Το θέμα είναι πώς θα γίνει η εφαρμογή. Γιατί αν το αφήσουμε open-ended, θα πρέπει να εξηγήσουμε πώς ο παράγοντας ε, σταθερότητας και ανάπτυξης ως προϋπόθεση θα συνδυαστεί με, την πολιτική του Ταμείου Συνοχής. Πάντως, πιστεύω ότι για να, να τη σημαντική αυτής πρότασης είναι να εξηγήσουμε τι σημαίνει η σύνδεση με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης αλλά και την ε, πολιτική συνοχή, την προσθέμενη αξία που προκύπτει από την πολιτική συνοχή. Και πολύ γενναία είναι η τροπολογία 44 που προτείνει διαγραφή ολόκληρης της προσέγγισης αυτής της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας. Είναι πολύ τολμηρή αυτή η προσέγγιση κατάργησης της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας και σας ε, ομολογώ ότι στην ομάδα μου δεν θα συμφωνήσουν όλοι οι ευρωβουλευτές. Πιστεύω ότι θα υπάρξει διάσταση απόψεων ε, και μεταξύ των φιλελευθέρων. Εγώ είμαι υπέρ, αλλά δεν μπορώ να σας εγγυηθώ ότι όλοι οι φιλελεύθεροι εστερνίζονται τη γνώμη μου. Και έρχομαι και σε ένα πολύ σοβαρό θέμα τώρα. Επειδή είμαι και μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών, έκανα αυτούς τους υπολογισμούς, όλους τους υπολογισμούς, και θα σας τους στείλω και στον κύριο Νίστερ και στους συνεισηγητές ε, και στα μέλη τους υπολογισμούς για τα διάφορα κονδύλια. Γιατί το κύριο πρόβλημα και στη συζητήση εδώ στο Κοινοβούλιο αλλά και στο Συμβούλιο θα είναι οι διαφορές μεταξύ των διαφόρων κονδυλίων και σε αυτές τις τρέχουσες δημοσιονομικές προοπτικές και στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο θα δείτε ότι υιοθέτησα τα στοιχεία και τους αριθμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα έλεγα λοιπόν πρώτα ότι δεν ευσταθεί το ότι τα κράτη-μέλη δεν είχαν μεθοδολογία για να υπολογίσουν τα κονδύλια για την επόμενη περίοδο. Όλα τα εθνικά υπουργεία και οι τοπικές αρχές έχουν ήδη κάνει τους υπολογισμούς τους με βάση τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής του περασμένου Ιουλίου και ξέρουν ε, τι κονδύλια θα πάρουν, αν είναι ε, μειονεκτικές περιοχές, σύγκλησης ή, καλα... ή ανεπτυγμένες περιοχές. Γνωρίζουν τι δικαιούνται με βάση την κατηγορία στην οποία ανήκουν. Και υπάρχει αυτή η μεθοδολογία. Ήταν διαθέσιμη στα κράτη-μέλη. Βέβαια αυτή η περιοχες γνωριζουν τι δικαιουνται με είναι διαφορετική από αυτή του ε, παραρτήματος 2, ε, παράγραφος 2 παράρτημα 1 του 1083 γιατί το 2 είναι το ανάτοτα όρια, το 3 είναι οι πολιτικές ε, μεταρρυθμίσεις και το 1 είναι οι προσαρμογές. Τώρα, φαίνεται ότι ίση μεταχείριση επιφυλάσσεται σε όλες τις περιφέρειες για τον υπολογισμό των κονδύλιων. Δεν υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις ανάλογα με το μέγεθος των χωρών ε, ή των περιφερειών. Βέβαια, αν κανείς δεν έχει όλα τα στοιχεία στην διάθεσή του, βρίσκεται σε αμηχανία, γιατί βλέπει ότι οι μεκτικές περιοχές θα έχουν 20% ε, λιγότερα κονδύλια και οι περιοχές συγκλήσει 47% λιγότερα. Αν κάνετε όμως κατά κεφαλή τους υπολογισμούς, θα δείτε ότι οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές θα λάβουν 6 ευρώ το χρόνο περισσότερο από ό,τι τώρα. Ενώ οι περισσότερο ανεπτυγμένες περιοχές θα λάβουν 0,8 ευρώ περισσότερα από ό,τι τώρα και οι μεταβατικές περιοχές είναι, γενικώ λαμβάνουν λιγότερα, είναι διαφορετικό το θέμα, θα πρέπει να γίνει ο υπολογισμός ε, της, του χαρακτηρισμού αυτού της μετάβασης. Πάντως, 17 περιοχές, 31 εκατομμύρια από τις περιοχές σύγκλησης θα πάνε στις μεταβατικές και 3 θα πάνε από, τις, από την κατηγορία σύγκλησης στις ενεπτυγμένες. Οπότε υπάρχουν πολλές αλλαγές. Και έρχομαι τώρα στη δική μου πρόταση. Τα κονδύλια υπολογίζονται με πολύ σωστό τρόπο. Το πρόβλημα με το κάπινγκ, το προσδιορισμό των ορίων, είναι σαφές. Έχουμε 0,51% ε, γενικώ, ακόμη και για το μέσο transit. Και αν έχουμε λιγότερο 0,51, ε, φυσικά και το κάπινγκ θα πρέπει να είναι χαμηλότερο. Και ερχόμαστε στη δική μου πρόταση τώρα, που δεν προκύπτει άμεσα από τον, από τον κανονισμό, αλλά επειδή έχουμε αυτά τα 11% ε, για διαπραγμάτευση, πιστεύω ότι είναι θεμελιώδη σημασία. Αν έχουμε μια μεγάλη χώρα και έχουμε, έχει αυτή περιοχές και στις τρεις κατηγορίες, μειονεκτικές, ε, μεταβατικές ε, και στις ανεπτυγμένες, η οικονομία είναι τόσο μεγάλη που με, το, με τη μείωση αυτή δεν θα έχει μεγάλη διαφορά στο συνολικό κονδύλιο. Αυτά για τις μεγάλες χώρες. Για τις μικρές όμως χώρες που δεν έχουν και πολύ καλές επιδόσεις και έχει η ΝΑΤΣ ε, μόνο σε μία περιοχή, τώρα η καταποκοπή του 051 θα μειώσει αισθητά το συνολικό κονδύλιο. Και υπάρχουν και κάποιες χώρες που έχουν μειονεκτικέ περιοχές στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο και θα πάρουν λιγότερο κατά 25% από τους τρέχοντα κονδύλια εξαιτία του κάπινγκ. Και φυσικά θα πρέπει να μειωθεί το κάπινγκ γιατί έχουμε λιγότερα κονδύλια, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει και κάτι άλλο που είναι απαράδεκτο. Το υπάρχον κάπινγκ, το ανώτατο όριο, ε, έχει, από 2,3 έχει περάσει το 2,7. Οπότε, αν έχουμε 57% του, του ΑΕΠ θα έχουμε 3,2 κάπινγκ. Ανάλογα με το ΑΕΠ υπολογίζεται και μειώνεται το κάπινγκ. Και στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο η Επιτροπή πρότεινε κατά αποκοπή 2,5% κάπινγκ για όλους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με, την, με το ελαστικό αυτό ποσοστό του κάπινγκ προτείνει και μία διάταξη που λέει ότι για να συνεχιστούν οι στόχοι το διαρθρωτικό ταμείο και να μειωθούν οι ανισότητες ε, στα κατακεφαλήν εισοδήματα, θα γίνει κατανομή του κάπινγκ, αυτού του του ορίου. Δεν ξέρω γιατί ε, ενώ αρχικά πρότεινε κάτι τέτοιο τελικά απέκλεινε από αυτή την προεσέγγιση. Περισσότερα κονδύλια δεν θα δοθούν. Το ξέρω αυτό από την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Πάντως το 2,5% να το μοιράσουμε, αυτό το 2,5% από 2,2 έως 2,7. Το κονδύλιο το συνολικό δεν θα, τροπο, θα τροποποιηθεί. Και είναι και πιο ελαστική η κατάσταση. Γιατί θα ισχύσουν οι αρχές της συνοχής σε τελική ανάλυση. Αν, κα... αν κάποιο κράτος δεν έχει καλές επιδόσεις, αν έχει καλή απορρόφηση, θα πρέπει και αυτό να ληφθεί υπόψη, αν δεν υπάρχει καλή απορρόφηση όχι. Αν όμως ε, βλέψουμε ένα καταποκοπή ανελαστικό 2,5% αντί να έχουμε ένα spread, μια ελαστικότητα, τότε πολλές χώρες θα χάσουν ε, πολύ σημαντικά κονδύλια. Διαφωνώ λοιπόν. Προτείνω ένα πιο ελαστικό κάπινγκ. Πάντως ευχαριστώ θερμά τους συγητές γιατί πραγματικά είναι πολύ γενναία και τολμηρή η πρότασή τους. Δεν ξέρω τελικά τι θα γίνει στις διαπραγματεύσεις. Πάντως πιστεύω ότι θα υπάρξει μεγάλη αντιπαράθεση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ειδικά αν επιμείνει στη θέση της. Πιστεύω ότι εμείς θα πρέπει να συμπληρωθούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να ενισχύσουμε τη θέση μας ώστε να μην ενδώσουμε προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Ελίζα Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρώτα τους εισηγητές. βλέπει κανείς και τη στρατηγική στην οποία βασίστηκαν. Ένα μέρος αυτής το συζητήσαμε στην ομάδα εργασίας και ιδίω του κοινού στρατηγικού πλαισίου κοινού πλαισίου στρατηγικής. Εγώ προσωπικά έχω κάποιες αμφιβολίες. Άλλωστε δεν έχω καταλήξει ακόμη. Εάν δηλαδή είναι πραγματικά καλό το στρατηγικό πλαίσιο να λάβει τόσο υψηλή αξία ώστε να μπει στον κανονισμό. Διότι τότε το καταγράφουμε πια πάρα πολύ στέρεα. Εμείς εγκαταλείπουμε τότε δηλαδή την ευκαμψία για τα 7 χρόνια. Εγώ θα προτιμούσα να επινοήσουμε μια διαδικασία που να την εγγράψουμε στον κανονισμό για το τι θα κάνουμε. Τι θα το κάνουμε αυτό το στρατηγικό πλαίσιο. Ποια θα είναι η διαδικασία δηλαδή μεταξύ Κοινοβουλίου και Κομισιόν για να υπάρχει ένα εργαλείο ευκαμψίας για αυτά τα 7 χρόνια για το στρατηγικό πλαίσιο. Γιατί δεν ξέρουμε σε 7 χρόνια τι μας περιμένει. και όταν κάναμε τον άλλο κανονισμό δεν είχαμε ιδέα τι θα σημάνει η κρίση και ποια μέτρα θα καταστούν απαραίτητα. Και γι' αυτό θέλω να το ξανασκεφτούμε. Αν θα το βάλουμε στο παράρτημα και επομένω στο νομοθετικό κείμενο. Αν αυτό δηλαδή είναι καλή ιδέα. Εγώ είμαι ανοιχτή απέναντι στα επιχειρήματά σα, αλλά διατηρώ κάποιε επιφυλάξει. Το δεύτερο που μου φαίνεται ενδιαφέρον στις προτάσεις είναι τα σχετικά με το άρθρο 87, δηλαδή πώς θα, ποιος θα γίνει το πρόγραμμα. Εκεί η πρόταση της Κομισιόν ήταν πολύ αυστηρή. Δηλαδή δεν μπορούσε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη πολιτική επιτόπου. στην ουσία ήταν σταχυολογημένα τα προγράμματα και ταυτόχρονα και γραφειοκρατικά. Βλέπω λοιπόν τώρα ότι ο Λάμπερτ και η Κωνσταντσε έκαναν σοβαρή προσπάθεια να εξεύρουν κάποιες λύσεις. Βλέπω ακόμη ότι προσπάθησαν να βάλουν κάποιους άξονες προτεραιοτήτων, που είναι καλή ιδέα. Νομίζω ωστόσο ότι δεν έχουν καταγραφεί όλα τα προβλήματα πρέπει να συζητήσουμε κι άλλο στην κατεύθυνση αυτή. Γνωρίζουμε ότι αυτοί οι άξονε προτεραιοτήτων είναι στην ουσία το κλειδί ολόκληρου του κανονισμού. Το ερώτημα είναι εάν θα το διατηρήσουμε το κλειδί αυτό για όλα ή αν θα σκεφτούμε αν μπορούμε να βάλουμε και κάποια ευκαμψία παραπάνω, κάποια flexibility ακόμα. Στις προτάσεις των δύο εισηγητών φαίνεται όλοι οι άξονες προτεραιότητα να πάνε σε μια κατεύθυνση. Η ευκαμψία δηλαδή να αναφέρεται στα ταμεία, στις περιφέρειες, να είναι αυτό ο προγραμματισμός αλλά πιο light, ένας άξονας προτεραιότητα να οδηγεί σε ένα στόχο, εγώ έτσι κατάλαβα από αυτά που είπατε τουλάχιστον, αλλά και πλήρωνες άξονες μπορούν να οδηγούν σε ένα στόχο. Αλλά μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σημαίνει όχι μονάχα όλοι οι άξονες να οδηγούν στον ίδιο στόχο, αλλά να εξετάζει κανείς και πώς μπορεί να γίνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Όπως για παράδειγμα για τα ITI ή για τις Local Development Groups. Και νομίζω ότι εκεί ακόμα δεν έχετε βρει τις λύσεις και πρέπει να συζητηθεί κι άλλο. Τώρα, η διαγραφή του αποθεματικού επιδότησης εμένα μου φαίνεται λάθος. Εγώ προτείνω να διαγραφούν οι κυρώσεις και να διατηρηθεί το θετικό μέρος. γιατί αυτό θα συμβάλλει στην καλύτερη αποδοτικότητα των προγραμμάτων. Αυτό που βρίσκω προβληματικό είναι η αποδυνάμωση των ε, συμβάσεων εταιρικής σχέσης αυτό ο αυτή η πολύ γενική διατύπωση με αυτή την cross-reference στην ε, παράγραφο α. Εγώ θυμάμαι νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό είναι κρίμα να διαγραφούν ορισμένα στοιχεία και εμείς ε, δεν θα συμφωνήσουμε. Τώρα, για το πώς εφαρμόζεται η εταιρική σχέση, εγώ βρίσκω ότι εδώ αποδυναμώνεται ταυτόχρονα, αλλά και μπορούμε να το συζητήσουμε βέβαια αυτό, μήπως επιλέξουμε άλλη διατύπωση, εγώ θεωρώ πάντως ότι αποδυναμώνεται, ταυτόχρονα γίνεται μία παραπομπή στο 5, αν όμως αποδυναμωθεί η σύμβαση εταιρικής σχέσης, τότε δεν διευκολύνουν καν οι παραπομπές αυτές. Οι οριζόντιες παραπομπές. Τώρα, αυτά είναι τα πιο βασικά, διότι έχω και πολλές τροπολογίες οι οποίες στρέφονται ακριβώς γύρω από αυτούς τους τομείς και πρέπει να βρούμε κάποιες κοινέ λύσεις. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε όλα όσα λέτε ακριβώς. Αλλά αυτός ο στρατηγικός σας προβληματισμός και η προσπάθεια απλούστευσης μας βρίσκει σύμφωνες αλλά νομίζω ότι χωρούν και κάποιες βελτιώσεις. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ο Βλάσακ δεν είναι εδώ. έχεις το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο κύριος Ομαρτζή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές και όσους τους βοήθησαν για την ε, εργασία την οποία μας παρουσίασαν. Η ομάδα μας θα καταθέσει συμπληρωματικές τροπολογίες στην έκθεση που έχει παρουσιαστεί. Θα ήθελα όμως να πω ότι σε γενικές γραμμές συμφωνούμε με την πρώτη σειρά αυτή των τροπολογιών και όπως είπε ο συνάδελφος Βαν έχει μεγάλη σημασία να υπογραμμίσουμε τις πολιτικές θέσεις τις οποίες θα καταλήξει η Επιτροπή μας. Στόχος τους είναι ο σεβασμός μιας κάποια σειρά αρχών στις οποίες έχουμε καταλήξει απαραίτητον για την περιφερειακή πολιτική. Έχω όμως την αίσθηση ότι το κείμενο το οποίο μας προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εν πολλής αντίστοιχο με την στρατηγική ε, για το 2020. Η στρατηγική 2020 είναι μια μακροοικονομική στρατηγική αναπτυγμένη για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορεί να εφαρμοστεί ως έχει στις περιφέρειες. Οι περιφέρειες έχουν ανάγκη από μια κάποια στήριξη η οποία θα τις βοηθήσει να διατυπώσουν τη δική τους πρόταση για τη στρατηγική τους ανάπτυξη. Πέρα από αυτό θα συμφωνήσω με τις προτάσεις των εισηγητών για να καταργηθεί η λεγόμενη μακροοικονομική αιρεσιμότητα θα πρέπει περισσότερες αποφάσεις ε, που λαμβάνονται σε επίπεδο κρατών μελών να καλύπτουν τις ανάγκες των περιφερειών, αλλά δεν θα πρέπει οι περιφερειές να πληρώνουν το τίμημα των προβληματικών αποφάσεων που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, μόνο και μόνο για να επανέλθουν σε μια δημοσιονομική ισορροπία. Γι' αυτό λοιπόν η Επιτροπή μας, ε, ομόφωνα σχεδόν από ό,τι βλέπω, ε, δεν θα δεχθεί αυτό το αποθεματικό επίδοσης. Σχετικά τώρα με την εκ των προτέρων προϋπόθεση. Εδώ η Επιτροπή μας θα πρέπει να καταθέσει κάποιες τροπολογίες και στα παραρτήματα, ιδιαίτερα στο παράρτημα υπαριθμού 4, το οποίο αναφέρεται λεπτομερώς στις συγκεκριμένες αυτές προϋποθέσεις. Γιατί μάλιστα κάποιες από τις προϋποθέσεις αυτές έχουν ξεπεραστεί πλέον από το ίδιο το πλαίσιο εφαρμογής των οδηγιών στις οποίες αναφέρεται για τις ε, προϋποθέσεις οι οποίες ανήκουν στα κράτη-μέλη, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο άρθρο 14. Εμείς θα θέλαμε να καταργηθεί κάτι το οποίο ε, τίνει να επιβληθεί στις περιφέρειες και που προέρχεται από την λεγόμενη διαδικασία των ευρωπαϊκών εξαμήνων. Να αναφερθώ τώρα και στις πλέον απόμακρες περιοχές σχετικά με, το ειδικό με την ειδική δημοσιονομική πρόβλεψη για τις περιφέρειες αυτές. Οι γνώμες είναι γνωστές και ελπίζω και η γνώμη της Επιτροπής μας να αντικατοπτρίζεται στην δεύτερη σειρά των τροπολογιών. Η τροπολογία αυτή για αυτές τις απόμακρες περιοχές θα πρέπει να επανισάγει τα ελάχιστα ποσά, τα ελάχιστα ποσοστά, όπως είχε προβλεφθεί στο παρελθόν. Προσωπικά εγώ δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει απόκληση από αυτή την αρχή. Ίσως έχω και κάποιες άλλες λεπτομέρειες τις οποίες θα αναφέρω προχωρώντας τη συζήτηση. Θα κλείσω λέγοντας ότι η επεξεργασία της εταιρική αυτής σύμβασης κάθε φορά θα πρέπει να γίνεται από το κράτο μέλος και τις περιφερειακές αρχές εν πλήρη διαβουλεύση και όχι μόνο από το κράτος μόνο του μετά από απλή διαβούλευση ε, των υπολείπων εταίρων. Αυτό είναι κάτι το οποίο εξασθενεί αν θέλετε τη διαδικασία. Και μια τελευταία παρατήρηση ελπίζω τις θέσεις ε, των εισηγητών να τις υποστηρίξουμε καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας πλήρως να έχουμε μια σκληρή θα έλεγα στάση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Uh, uh, Ευχαριστώ. Όλμπρεχτ είναι ο πρώτος ομιλητής. yes, Θα συνεχίσω αγγλικά γιατί το κείμενο όπως είπα το αρχικό ήταν στα αγγλικά. Πρώτον, Μόλις ε, ξεκινήσαμε τώρα την τελική φάση της προσπάθειας την οποία κάνουμε, θέλω να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές. Υπάρχουν αρκετά στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά. Συμφωνώ με την Κρόλη η οποία λέει ότι ο κανονισμός αυτός είναι η βάση όλων των υπολείπων επιμέρους κανονισμών. Και η απόφαση την οποία θα πάρουμε για το Γενικό Κανονισμό σαφώς και θα χαρακτηρίσει τις θέσεις του Κοινοβουλίου για το υπόλοιπο πακέτο, για το σύνολο του πακέτου των κανονισμών. Κάποιες από τις αποφάσεις αυτές που υποτίθεται είναι γενικής φύσεως, στην ουσία θα είναι αποφασιστικές για όλους τους υπόλοιπους ε, κανονισμούς και όλα τα υπόλοιπα ταμεία. Κάποιες παρατηρήσεις τώρα επιμέρους. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία Uh, this is crucial element because, uh, uh, as we know, we have today, we have the proposal. Σχετικά με το κοινό στρατηγικό πλαίσιο υπάρχει μια πρόταση για ένα κοινό πρόγραμμα για πέντε ταμεία. Υπάρχει ένας γενικός κανονισμός σε δύο τμήματα. Το πρώτο είναι, το πρώτο είναι όλα τα υπόλοιπα εκτός από τη συνοχή και το δεύτερο είναι μόνο η συνοχή. Τα τέσσερα λοιπόν το πρώτο και ε, το δεύτερο είναι ποιο είναι το καθεστώς του κανονισμού αυτού. Μιλάμε για ένα απλό κανονισμό ή μιλάμε για πρόταση κανονισμού ή μιλάμε για ένα λειτουργικό κείμενο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξ αρχής έχει προτείνει επίσης την διαδικασία των κατεξουσιοδότηση πράξεων. Και βρισκόμαστε σε μια ξεκάθαρη τώρα κατάσταση. Το κείμενο εργασίας, το οποίο προτείνεται στη φάση αυτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει ένα χαρακτήρα τέτοιο έτσι ώστε δεν μπορεί να θεωρηθεί νομικά δεσμευτικό. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχει αποδείξει αυτό με το κείμενό της. Η αντίδρασή μας σε αυτό μπορεί να πάει προς δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, να συμφωνήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να πούμε ότι πράγματι το κείμενο αυτό δεν μπορεί να καταστεί νομικά δεσμευτικό. Είναι ένα ενημερωτικό κείμενο, είναι κάποιες κατευθυντήριες γραμμές και να συμφωνήσουμε μαζί της. Οπότε σε αυτή τη διαδικασία τα πράγματα θα προχωρήσουν. Ή να δεχτούμε την πρόταση των εισηγητών. Να πούμε ότι ας πάρουμε τα θέματα προς συζήτηση, αλλά ας βάλουμε διαφορετικό περιεχόμενο και ας το καταστήσουμε το κείμενο νομικά δεσμευτικό, νομικά ισχυρό. Κρατάμε το όνομα λοιπόν και βάζουμε ένα διαφορετικό περιεχόμενο στο όνομα αυτό δίνοντας την δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας εξηγήσει πώς νομικά θα καταστήσει τα πέντε αυτά τα ταμεία συμπληρωματικά και πώς θα μετατρέψει τον κοινό προγραμματισμό σε πρακτική εφαρμογή. Αυτός είναι ο στόχος τον οποίο θέλουμε να πετύχουμε. Δεν θα τον πετύχουμε πάρα πολύ γρήγορα βέβαια, γιατί όσο συζητάμε την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση τόσο πιο επιμέρους αναγκαστικά θέματα μας απασχολούν. Παρ' όλα αυτά την προσπάθεια θα πρέπει να την κάνουμε. Ο μοναδικός τρόπος λοιπόν αντίδρασης από πλευράς μας είναι να υπάρξει ένα νέο κείμενο. Αυτό έχει απόλυτη λογική. Είναι ενδιαφέρον τώρα να πούμε ότι το κείμενο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ιδιαίτερο χρήσιμο, αλλά όχι σαν νομικό κείμενο, αλλά σαν κατευθυντήριες γραμμές. να πω κάτι ανεπίσημα. Στην ουσία η Επιτροπή φταίει για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Μας είχε υποσχεθεί συγκεκριμένες κομβικές δράσεις στα πλαίσια του στρατηγικού αυτού πακέτου και τώρα εδώ μας παρουσιάζει κάποιες γενικές προτεραιότητες. Συνεπώς λοιπόν έχουμε δύο διαφορετικά επίπεδα λειτουργικών κειμένων εδώ ξεχωριστά το ένα από το άλλο. Θα πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά όχι σαν νομικό κείμενο. Δεύτερη παρατήρηση. Θα υποστηρίξω την ιδέα ότι το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί σαν παράδειγμα αλλά λαμβάνοντας υπόψη το χαρακτήρα συμπληρωματικότητας των ταμείων. Και πιστεύω ότι όταν έχουμε ένα νομικό κείμενο, συνέπεια θα είναι να αναγνωρίσουμε πλέον μια πολλαπλή ύπαρξη των συγκεκριμένων ταμείων και ξεχωριστούς τρόπους λειτουργίας. Τώρα για το πώς θα συνάπτονται οι συμφωνίες αυτές, οι εταιρικέ συμφωνίες, οι συμβάσεις, δεν θα αναφερθούμε στα θέματα του κώδικα συμπεριφοράς που ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητα όταν συζητιούνται ανάμεσα στα κράτη. Η πρόταση που γίνεται είναι να κερδίσουμε χρόνο ουσιαστικά. Το θέμα δεν είναι όμως μόνο αυτό. Αν κατάλαβα καλά τους εισηγητές, αυτό το οποίο θέλουν είναι μια σταδιακή αντιμετώπιση. Πρώτο, να ασχοληθούμε με τα συμβόλαια αυτά τα, της εταιρικότητας και αυτή τη στιγμή υπογραφούν τότε να περνάμε στα λειτουργικά προγράμματα μετά σε μια δεύτερη φάση. Αυτό τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε με τα δύο αυτά επίπεδα να ασχοληθούμε ταυτόχρονα. Απλά η στάση, η στάση μας απέναντί τους θα πρέπει να είναι σε φάση. Στην πρώτη φάση η υπογραφή των συμβάσεων, στη δεύτερη φάση η κατάθεση των λειτουργικών προγραμμάτων. Έτσι εμείς ενισχύουμε το ρόλο αυτών των προγραμμάτων. Και κάποιες ε, λιγότερο ίσως σημαντικές παρατηρήσεις να μου επιτρέψετε να κάνω. Θα ήθελα να ζητήσω από τους εισηγητές τι εννοούν όταν ε, συζητούν τα χρηματοδοτικά μέσα και αναφέρονται σε θεματολογικούς στόχους και συγκεκριμένους στόχους. Καταλαβαίνω, θεματικούς ή θεματολογικούς στόχους το καταλαβαίνω. Συγκεκριμένους επιμέρους στόχους δεν το καταλαβαίνω. Τι εννοούν εδώ. Έχουμε επίσης ένα θέμα και με το 17. Στις τροπολογίες σας προτείνετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί τις πληροφορίες που συλλέγει πριν να μπορεί να έχει τη δυνατότητα να υιοθετήσει ένα πρόγραμμα το οποίο να διακόπτει την πληρωμή συγκεκριμένων προγραμμάτων επί τη βάση των κανόνων των συγκεκριμένων. Γιατί στο Περιφερειακό Ταμείο, σαν παράδειγμα, δεν υπάρχουν κανόνες ξεκάθαροι σε σχέση με τη διακοπή των πληρωμών. Ξέρω ότι στο Ταμείο Σύνοχης, σύμφωνα με τη συνθήκη ε, του Μάστριχτ, υπάρχουν κανόνες σχετικά με τη διακοπή πληρωμών, αλλά στο περιφερειακό δεν υπάρχουν, όπως και ίσως και σε άλλα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διευκρινίσουμε. Σας ευχαριστώ που εισάγετε και το θέμα του καταλόγου των κριτηρίων. Ε, μπορούμε εδώ να ξεχωρίσουμε τις περιοχές καλύτερα, να μιλήσουμε για αστικές περιοχές, περιοχές αστικών συγκεντρώσεων. Αυτά είναι λεπτομέρειες στα οποία θα έρθουμε. Ευχαριστώ. Ernst. Ja, recht vielen Dank. Es ist schon viel Lobenswertes gesagt worden äh, zu dem, was Λέχθηκαν πολλά για τα όσα έχουν υποβάλει οι ε, εισηγητέ. Μπορώ να συμφωνήσω σε πολλά για τη, μακροοικονομικά, ε, για τη μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Σωστό να διαγραφεί το ίδιο το αποθεματικό επίδοσης και μια παράγραφος ακόμη που διαλαμβάνει την βασική ιδέα και κάπου τη διατηρεί της ε, επίδοσης, δηλαδή Εκεί με βρίσκει σύμφωνη. Για το 46 περισσότερο χρόνο δηλαδή για τα προγράμματα νομίζω ότι εδώ είναι καλή η πρόταση και μπορεί να τη δεχτεί κανείς. Προσωπικά με ενδιαφέρει η συμπερίληψη του δημογραφικού παράγοντα, κάτι το οποίο εμάς ε, μας φαίνεται πολύ σημαντικό. Και η αναφορά στην, ε, στον ΦΠΑ. Τώρα, για την μακροοικονομική, μη μάλλον για την ex ante conditionality για την εξάντη conditionality και πρέπει να συζητηθεί. Αντιλαμβάνομαι τι θέλετε και το βρίσκω σωστό σε σχέση δηλαδή με την πολιτική συνοχή. Ότι αυτοί, αυτοί, οι όροι, αυτές οι αιρεσιμότητες πρέπει να παίζουν ρόλο. Αλλά πώς θα διατυπωθεί ή μήπως πρέπει η πρόταση να προσεγγιστεί τελείως διαφορετικά. Δηλαδή να πούν πώς θα πρέπει να είναι και πώς δεν θα πρέπει να είναι κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή να γίνει μια διάκριση, μια διαφοροποίηση μέσα στις προτάσεις που έχει κάνει η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω δηλαδή ότι με την διατύπωση αυτή πρέπει να την ξανασυζητήσουμε. Δεν τη βρίσκω να είναι συνεπής. Τώρα η αστική διάσταση και οι λίστες αστικών κέντρων. Τι λίστες είναι αυτές κριτηρίων, αυτό χρειάζεται λίγη συζήτηση ακόμη. Είμαι επιφυλακτική, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να ε, αντιληφθεί ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Τώρα, άξονε προτεραιοτήτων και η διασύνδεση με τους στόχους. Αυτά τα είπε η κυρία Σρέντερ και με βρίσκει σύμφωνη. Θεωρώ και εγώ λοιπόν ότι χρειάζεται παραπέρα συζήτηση. Κατά τα άλλα νομίζω στη δεύτερη δόση θα ακούσουμε και άλλα πράγματα για απογραφειοκρατικοποίηση και ούτω καθεξής. Τελευταίο τώρα τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει δηλαδή τι ακριβώς θέλουμε σε σχέση με τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τι ακριβώς δηλαδή εννοούμε. Εκεί νομίζω πρέπει να εγκύψουμε περισσότερο και να κάνουμε ακριβέστερες διατυπώσεις. Κατά τα λοιπά νομίζω, όπως είπα, ότι είναι καλή δουλειά και αποτελεί μια βάση και για περαιτέρω εργασία. Ευχαριστώ. Βλαντίμιρ. Μάνικα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή είναι η παρθενική μου ομιλία στην Επιτροπή Είναι, ήμουν μέλος προηγουμένως στην Επιτροπή Προϋπολογισμών για 8 χρόνια, 8 ολόκληρα χρόνια και μάλιστα ήμουν και ο εισηγητής για τον προϋπολογισμό του 2010. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τους συνεισηγητές για το αξιόλογο έργο τους. Πιστεύω ότι αυτό το έγγραφο θα γίνει μια πολύ καλή βάση και για το μελλοντικό μας ε, έργο και τις συζητήσεις. Πριν από μερικά χρόνια, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετείχαν σε μια συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και είπαν ότι θα πρέπει να μειωθούν τα κονδύλια για τα κράτη-μέλη κατά 10% εξαιτίας της χαμηλής ε, απορρόφησης. Τότε μάλιστα ήμουν δήμαρχος μιας πόλης και είχα και εμπειρία από πρώτο χέρι για το θέμα αυτό που με δίδαξε ότι χρειάστηκαν διετή συζητήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εκταμιευθούν κονδύλια εξαιτίας της ε, υπερβολικής γραφειοκρατίας. Μετά από επίσκεψη όμως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και τη συζήτηση που έγινε, καταφέραμε να περιορίσουμε, να πλουστεύσουμε τη γραφειοκρατία, να περιορίσουμε τις γραφειοκρατικές διατυπώσεις, το ελάχιστο, αλλά έγινε μια μεταφορά της γραφειοκρατίας προς τα κράτη-μέλη, γιατί υπάρχει διαφορετική η γραφειοκρατία που ισχύει σε κάθε κράτος, διαφορετικοί είναι οι ισχύοντες κανόνες και πιστεύω ότι η προσπάθεια να μειωθεί το γραφειοκρατικό άκθος θα πρέπει να γίνεται σε όλα τα κράτη-μέλη προκειμένου να καταλήξουμε σε μια εναρμόνιση τελικά. Ο κύριος Γκουτμάνης στη δήλωση που μας έκανε είπε ότι μια χώρα είναι υπερβολικά καλή στην, απο... απορρόφηση ή κάπως οκνηρή. Νομίζω ότι όμως αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο είναι ποιοι είναι ισχύοντες κανόνες για την απορρόφηση. Εγώ είμαι αρμόδιος για μια μεγάλη περιφέρεια της Ευρωπαϊκής και ξέρω ότι κάποιες χώρες έχουν αδυναμίες στην υποδομή τους. Γι' αυτό και μερικές φορές καλούνται να υπερκεράσουν τεράστια εμπόδια εξαιτίας των προβληματικών υποδομών. Για παράδειγμα, αν έχουμε μία πλημμύρα και δεν έχουμε αρκετές γέφυρες σε μία περιοχή, αμέσως επηρεάζεται το πρόγραμμα γιατί λαμβάνει κάποιο ε, κοινοτικά προγράμματα και κοινοτική χρηματοδότηση που προβλέπουν όμως συγχρηματοδότηση από μια χώρα. Βέβαια, όταν ε, έχουμε μια θεομηνία, μια πλημμύρα, θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις τρέχουσες συνθήκες. Και δημιουργούνται και απρόβλεπτες δαπάνες που δεν εμπίπτουν πια στις επιλέξιμε δαπάνε. Έτσι δημιουργείται πρόβλημα. Και πρόβλημα υπάρχει και από το πλαίσιο της χρηματοδότησης και από τους ε, ορισμούς και τους κανόνες που ισχύουν. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο ελαστικοί για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα που ανακύπτουν ευνίδια. Πάντως πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε πολύ καλούς κανόνες χάρη στη συνεργασία για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ευχαριστώ κύριο Σαλενκαρέκ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Κωνσταντς και τον Λάμπερτ για το έργο τους, γιατί πραγματικά είναι αξιέπαινο και ήδη είναι άξιοι συγχαρητηρίων, σε ό,τι αφορά τα σημεία σύγκλησης. Και εγώ θεωρώ ότι πραγματικά είναι απαραίτητο το κοινό στρατηγικό πλαίσιο να πάρει τη μορφή μιας κατεξουσιοδότηση πράξης. Θα πρέπει να αποτελέσει παράρτημα του γενικού προπολογισμού και άρα να εμπίπτει στη συναπόφαση. Είναι προφανές. Επίσης, ασθενίζομαι την πρόταση ε, της κατάργησης του αποθεματικού επίδοσης, γιατί δεν είναι καθόλου καλή η ιδέα του αποθεματικού επίδοσης. Σε ό,τι αφορά την εξάντε αιρεσιμότητα, θα διευκολύνει την ε, απορροφητικότητα των ε, ταμείων και την εκταμίευση, αλλά θα πρέπει να περιορίζεται στο πεδίο εφαρμογής των ταμείων. Γιατί ο κίνδυνο είναι να δημιουργήσει αιρεσιμότητα ένα επιπλέον και υπέρμετρο γραφειοκρατικό άχθος. Προσοχή λοιπόν, πάντως ως ιδέα είναι ενδιαφέρουσα. Από την αρχή, πολλοί συνάδελφοι τάχθηκαν υπέρ, όπως και εγώ, της μακροοικονομικής αιρεσιμότητα. Δεν είναι μυστικό. Πριν από λίγο όμω, η Κωνσταντς μα είπε ότι το μέτρο αυτό ίσω βλάψει τελικά και πλήξει τις ε, περιφέρειες ε, λόγω ενός δημοσιονομικού ελλείμματος ε, για το οποίο δεν είναι υπεύθυνε ίδιες αλλά η κεντρική κυβέρνηση. Πιστεύω ότι η πολιτική συνοχή δεν θα πρέπει να αποσυνδέεται από τη γενική προσπάθεια λιτότητας που προσπαθούμε από όλες τις χώρες, που επιδιώκουμε και απαιτούμε από όλες τις χώρες. Θα πρέπει να το σκεφτούμε και αυτό. Οι εισηγητές πρότειναν να διαγραφεί των παραγράφων 3 και 4 του 20 για την αναστολή των πληρωμών για τα προγράμματα που δεν κρίνονται ιδιαίτερα αποδοτικά κατά την ενδιάμεση περίοδο αξιολόγησης. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να διαφυλάξουμε την παράγραφο αυτή για να μην ε, ε, εκενώσουμε περιεχομένου τις ε, απαιτήσει μας για επιδόσεις που είναι σημαντικές. Ίσως χρειαστεί κάποια αναδιατύπωση της παραγράφου για να αποφύγουμε αυτόματη ή πολύ ριζική εφαρμογή των κυρώσεων. Ναι, με αυτή, είμαι υπέρ τη παραγράφου, αλλά με μεγαλύτερη ελαστικότητα. Τώρα, σε ό,τι αφορά του μηχανισμού συντονισμού με τι μακροπεριφέρειες, να ληφθούν υπόψη και επίση ε, χρειαζόμαστε και ένα μηχανισμό ε, ε επί, υποχρεωτικό, για τις ε, μακροπρόθεσμες στρατηγικές. Επίσης, χρειαζόμαστε ε, ολοκληρωμένα εδαφικά πολιτή προγράμματα για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της ε, μακροπεριφερειακής στρατηγικής. Αυτά προς το παρόν. Φυσικά θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε και να συνεχίσουμε τη συζήτηση με τους συνεισηγητές και τους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ταμάς Πορέμπα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να λάβω το λόγο. Σίγουρα Εδώ και μήνες ασχολούμαστε στην Επιτροπή Ρέγγι για τη μελλοντική μορφή που θα λάβει η πολιτική συνοχή και το έργο μας είναι πολύ σημαντικό και πολύ αξιόλογο. Βέβαια πρόσφατα διαπιστώσαμε ότι η οριστική μορφή της πολιτικής συνοχής δεν θα γίνεται εκτός στα πλαίσια του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι εργαζόμαστε κενό και χωρίς δημοσιονομικές βάσεις. Κάτι που θα ήταν απαραίτητο για να προετοιμάσουμε το έγγραφό μας. Πολλό δε μάλλον που η πολιτική συνοχής είναι πολύ εύκολος στόχος για τις χώρες που είναι καθαροί πληρωτές και ζητούν οικονομίες. Και οι τελευταίες πληροφορίες από το Λεξεβούργο μας ανησυχούν, ιδιαίτερα για τις προτάσεις των ανατάτων ορίων και τα, τις τα ποσοστά απορρόφησης. Η πρόταση για την περικοπή του προπολογισμού είναι πολύ ανησυχητική και φυσικά η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, καλό θα ήταν να ληφθεί υπόψη τη συζήτηση και οι προτεραιότητες της να εισακουστούν γιατί και το δικό μας έργο είναι πολύ σημαντικό. Επανέρχομαι τώρα στην έκθεση. Θα ήθελα και εγώ να επενέσω τους συνεισηγητές για το πολύ αξιόλογο έργο τους και για τις πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις τους πολύ σωστά ζητάτε διαγραφή της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας, πολύ σωστά προτείνατε το ΦΠΑ να έρθει υπόψη. Επίσης θα ήθελα να ασκήσουμε περισσότερη πίεση για να ενισχυθεί ο ρόλος της μακροοικονομικής στρατηγικής των λειτουργικών προγραμμάτων και να τονίσουμε ότι η μακροπεριφερειακή στρατηγική και τα σχετικά λειτουργικά προγράμματα εξυπηρετούν την πολιτική συνοχή και την εξισορρόπηση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών και την συνολική ανάπτυξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ομάδα των μεταρρυθμιστών και συντηρητικών θα καταθέσει πρωτο... για το θέμα αυτό σε συνεργασία και συμφωνία με τους συνεισηγητές. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ε, την μείωση του ποσοστού απορρόφησης κατά στο 2,5% γιατί δεν θα βοηθήσουμε έτσι τις χώρες που έχουν χαμηλότερες επιδόσεις και που αγωνίζονται να ξεπεράσουν την ισχύουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Πάντως ευχαριστώ τους συνεισηγητές γιατί οι περισσότερες τροπολογίες βαίνουν προς την κατεύθυνση, λαμβάνουν υπόψη τις ευαισθησίες μας και θα συμβάλλουμε και εμείς με τις δικές μας τροπολογίες. Θα προσπαθήσουμε να προτείνουμε λύσεις που θα τύχουν ε, υποστήριξη της ε, Επιτροπής μας, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε ομόφωνη γνώμη. Ευχαριστώ. Η κυρία Μανέσκου. Ε, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ξεκινώντας θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Λάμπερτ και την Κωστός γιατί έχουν πολύ βελτιώσει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συμφωνώ και με τις προτάσεις τις οποίες έκαναν και δεν θα επαναλάβω πράγματα τα οποία ακούστηκαν αναλυτικά από τους προηγούμενους ομιλητές. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ λίγο στην εταιρική σχέση του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Στο άρθρο 54 σχετικά με τις προσοδοφόρες δράσεις νομίζω ότι εδώ δεν υπάρχει ουσιαστική αναφορά στη σχέση του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, διότι θεωρείται μια τέτοια σχέση ιδιαίτερως περίπλοκη. Υπάρχουν δύο τρόποι υπολογισμού των εσόδων και αυτό είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει μια νομική έλλειψη ασφαλείας. Θεωρώ ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε μια καλύτερη λύση και να εντοπίσουμε μια πιο σωστή μέθοδο υπολογισμού έτσι όπως προβλέπεται στο 54 1 α μικρό. Στο άρθρο 55 επίσης καλό θα ήταν να διευκρινιστεί ότι τα κριτήρια επιλεξιμότητας θα πρέπει να ισχύουν και για τα λεγόμενα PPP όπως επίσης και για τα συμβάσεις οι οποίες είναι κάτω από ε, διαχείριση του δημόσιου τομέα. Έτσι θα καλύψουμε και τα συμφέροντα του δημόσιου τομέα αλλά και τα συμφέροντα του ιδιωτικού, των επιχειρήσεων. Ένα άλλο θέμα το οποίο συνδέεται με τη διαφάνεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ζητήσει από τα κράτη-μέλη να καταθέσουν τα προγραμματικά τους κείμενα σε μία, σε μία ιστοσελίδα. Αυτό θα δημιουργήσει συνθήκες διαφανείας και θα επιτρέψει στον πολίτη να σχολιάσουν και να συνεισφέρουν τις προτάσεις τους σύμφωνα με αυτά τα οποία θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πολίτες λοιπόν μπορούν να συνεισφέρουν τελικά και πριν μάλιστα από την λήψη της τελικής απόφασης για ένα πρόγραμμα. Να παρατηρήσω επίσης ότι αυτό το οποίο υπογραμμίζεται εδώ είναι τα διάφορα μέσα ενημέρωσης, πληροφόρησης, κατάρτισης για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Όχι όμως για τον ιδιωτικό τομέα, όχι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Εάν πράγματι θέλουμε εμείς να είμαστε αποτελεσματικοί στα πλαίσια της στρατηγικής 2020 και για τον ιδιωτικό τομέα και για τις μικρομισές επιχειρήσεις, τότε θα πρέπει να προβλεφθούν και μέσα ενημέρωσης των συγκεκριμένων επιχειρήσεων και μάλιστα και μέσα όχι μόνο απλής ενημέρωσης αλλά και διαβούλευσης. Αυτό θα καταστήσει, θα έλεγα, τον διάλογο πιο αποτελεσματικό και θα φέρει σε στενότερη επαφή και συνεργασία τον ιδιωτικό τομέα με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Τώρα για τις, ε, αυτές τις εταιρικές συμβάσεις είναι σωστό αυτό το οποίο προτείνεται από τους δύο εισηγητές με την αντικατάσταση της, της περίοδου τριών μηνών από μια αντίστοιχη εξαμηνιαία. Νομίζω ότι αυτό είναι χρήσιμο. Ταυτόχρονα όμως θεωρώ ότι έχει μεγάλη σημασία να επιβάλλουμε στα κράτη-μέλη την υποχρέωση να διαβουλεύονται με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές. Είναι κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει επανειλημμένα. Θα πρέπει να υπάρξει μια διακυβέρνηση, αν θέλετε αυτή, της διαδικασίας αυτής με πολλούς εταίρους και η αγγλική λέξη shall θα πρέπει να αντικατασταθεί από την αγγλική λέξη must. Δηλαδή πρέπει να είναι υποχρεωμένες οι κεντρικές αρχές να διαβουλεύονται με τις περιφερειακές αρχές. Γιατί αλλιώς στην ουσία οι κυβερνήσεις, οι κεντρικές τα διαλέγουν κατά περίπτωση αν θα έλθουν σε επαφή ή δεν θα έλθουν σε επαφή. Να χαιρετήσω επίσης και την πρόταση των εισηγητών να καταργηθεί η παράγραφος η σχετική με τη μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Όπως είπε ο κύριος Γκοντμάνης, η ομάδα των φιλελευθέρων δεν υποστηρίζει την κατάργηση αυτής της μακροαιρεσιμότητας. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ο τρόπος με τον οποίο θα καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις. Θεωρώ ότι το μήνυμα το οποίο εστάλει από το Λουξεμβούργο από τις 13 χώρες, οι οποίες ε, είπαν ότι είναι κατά αυτής της ερεσιμότητας, είναι ξεκάθαρο. Αγαπητοί, ε, δεν θέλω βέβαια να περιοριστώ τον χρόνο αγόρευσή σας, γιατί είναι πολύ σημαντικό να διεξαχθεί σε βάθος συζήτηση, να μπορέσετε όλοι να αναπτύξετε τις θέσεις σας, αλλά περνάει η ώρα βέβαια. Αν μπορείτε λοιπόν να περιοριστείτε κάπως ο κ. Χρυσόγελος. Ευχαριστώ πολύ. Ε, η, η, έκθεση είναι ιδιαίτερα σημαντική και νομίζω θα είναι χρήσιμη και για τη συζήτηση και για προστίκη ορισμένων συμπληρωματικών ε, ορισμένων ε, τροποποιήσεων. Θα ήθελα να πω ότι συμφωνούμε να διαγραφεί διάταξη περί δημοσιονομικής ε, τιμωρίας στην πραγματικότητα, ερεσιμότητας γιατί ε, χρειάζονται θετικά κίνητρα και εργαλεία για να ενδυναμώσει η ικανότητα των περιφερειών και των τοπικών αρχών στο σχεδιασμό, στην ε, υλοποίηση και στην παρακολούθηση εξελόγηση των προγραμμάτων. Η τιμωρία δεν βοηθάει τίποτα, ούτε η απειλή τη τιμωρία από μόνη τη αρκεί. Το δεύτερο νομίζω που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ισχυρή διατύπωση στο κείμενο για να συμμετέχουν οι περιφέρειες στα σχέδια που αφορούν την περιοχή τους. Η ευχή έχουμε δει ότι δεν λειτουργεί και έχουμε την εμπειρία και από ε, διάφορα κράτη-μέλη. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει η δέσμευση για συναπόφαση των περιφερειών, για προετοιμασία των περιφερειών στο επίπεδο του σχεδιασμού, για συμμετοχή τους στην εταιρική ε, σύμβαση και στην αξιολόγηση και παρακολούθηση των προγραμμάτων. Και νομίζω αυτό πρέπει να μπει είτε στο γενικό κανονισμό που θα είναι ακόμα πιο ισχυρή δέσμευση, είτε τουλάχιστον στον, ε, στον ε, κώδικα ε, συμπεριφορά, στο Code of Conduct. Δεν νομίζω ότι πρέπει να αρκεστούμε στο θέμα σάλ ή ευχή. Ε, και η εμπειρία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δείχνει ότι όταν μπήκε το Κοινοβούλιο σε αυτή τη δικασία συναπόφαση, αυτό βελτίωσε όλη τη δικασία λήψη αποφάσεων. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να γίνει και στο επίπεδο των, των προγραμμάτων αυτών που συζητάμε είναι σημαντικό ότι εδώ πέρα συζητάμε για ταμεία τα οποία θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά πρέπει να πάμε και από την άλλη πλευρά και να βοηθήσουμε και τις χώρες και τις περιφέρειες να έχουν μια αντίστοιχη προσέγγιση συμπληρωματικότητα. Δηλαδή, όταν κάνουν το σχεδιασμό του, να αντιλαμβάνονται το σύνολο των δυνατοτήτων ε, και να λειτουργούν και αυτοί με την έννοια τη συμπληρωματικότητα των διαφόρων πηγών χρηματοδότηση. Να μην προσανατολίζεται μόνο στην υλοποίηση ορισμένων προγραμμάτων απασπασματικά. Ε, θα έλεγα ότι το Ταμείο επι, ίσω ε, Επιβράβευσης ίσως θα είχε ένα ενδιαφέρον και το αποθυματικό επίδοση θα έχει ενδιαφέρον αν καθορίσουμε τα κριτήρια. Αν δεν είναι μόνο κριτήρια οικονομικά, ίσω έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή αν μια περιφέρεια πετυχαίνει στόχους όπως είναι το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης, ίσως θα έχει ενδιαφέρον. Αν πετυχαίνει στόχους που συνδυάζει περιβαλλοντικά αποτελέσματα και ε, κοινωνική συνοχή, ίσως αυτό έχει σημασία να υπάρχει ένα αποθεματικό επίδοσης, αλλά που δεν είναι απλώς με οικονομικούς όρους. Δεν είναι δηλαδή ότι πέτυχε να απορροφήσει πόρους, αλλά πέτυχε στους στόχους που θέτουμε για έξυπνη, ε, αηφορική και ε, ε, ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή. Άρα λοιπόν ίσως έχει ενδιαφέρον. Και ήθελα να καταλήξω λέγοντας ότι έχω μία ανησυχία την οποία έχω διατυπώσει και ε, στη συζήτηση που κάνουμε για την κοινωνική συνοχή αλλά νομίζω ότι είναι κατάλληλο για εδώ. Είναι τα κριτήρια επιλεξιμότητας των περιφερειών και των χωρών ε, στα διαφορετικά ταμεία και στα ταμεία Συνοχής. Με βάση το άρθρο 82 του Γενικού Κανονισμού τα στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2006-2008 θα καθορίσουν την κατάταξη των περιφερειών και τα στατιστικά στοιχεία της περίοδου 2007-2009 για το Ταμείο Συνοχής. Όμως εδώ έχει επέλθει μια σημαντική αλλαγή λόγω της μεγάλης κρίσης και των μέτρων λιτότητας που έχουν οδηγήσει σε τεράστια ύφεση και σε αλλαγή της κατάστασης σε πολλές περιφέρειες. Άρα θα πρέπει να το δούμε στο γενικό κανονισμό πώς θα ενσωματώσουμε πιο πρόσφατα στοιχεία, τουλάχιστον μέχρι το 2011, να ενσωματώσουμε δηλαδή την περίοδο της κρίσης. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μιλήσουμε πραγματικά για περιφερειακή ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να τονίσω ε, στο επίπεδο του γενικού κανονισμού, αλλά και να το λάβουμε υπόψη και στα άλλα επιμέρου συζητήσει και τα άλλα ταμεία. Thank you very much, ε, Victor Ευχαριστώ κύριε Βίκτορ Μποστινάρο. Και εγώ ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φυσικά υποστηρίζω και καλωσορίζω και τη φιλοσοφία του Γενικού Κανονισμού και τις τροπολογίες των δύο αξιότιμων συνεισηγητών. Είναι πολύ σημαντική αυτή η προσπάθεια γιατί δείχνει πώς ε, με στενή συνεργασία μπορούμε όλες οι πολιτικές παρατάξεις να δημιουργήσουμε μία σμεστή και στεναρή έκθεση που θα μας βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Για μένα είναι πολύ θετικό αυτό και πολύ αξιόλογο. Δεύτερον, στι στις εταιρικές συμβάσεις και στον διοντολογικό κώδικα, τον κώδικα συμπεριφοράς, θα ήθελα να ενισχύσουμε τη θεσμική και διοικητική ικανότητα των κρατών μελών. Και αυτό είναι σημαντικό όχι γιατί μόνο μερικά αντιμετωπίζουν σήμερα τεράστια προβλήματα, αλλά με τη νέα ε, πολυσύνθετη περίπλοκη πολιτική συνοχής είναι σημαντικό να έχουμε ε, πολύ καλό επίπεδο θεσμικής ε, και διοικητικής ικανότητας για να έχουμε καλύτερη εφαρμογή και κατά κάποιο τρόπο να είναι υποχρεωμένα τα κράτη-μέλη να έχουν εύρυθμη διοίκηση και γι' αυτό θα πρέπει να την αναφέρουμε στις εταιρικές συμβάσεις και να προβλέψουμε και σημαντικούς αυστηρούς δεσμευτικούς κανόνες στον κώδικα συμπεριφοράς. Βέβαια θα δυσαρεστήσει μια τέτοια πρόταση κάποια κρατημέλη, αλλά για την καλύτερη εφαρμογή της πολιτικής συνοχής και θέλουμε καλύτερα αποτελέσματα και πιο ορατά και απτά της πολιτικής συνοχής, μόνο έτσι θα καταφέρουμε να ανατρέψουμε μια τάση που μέχρι στιγμής δεν είναι και πολύ θετική. Τώρα, η διευκόλυνση του Connecting Europe, το μέσο Connecting Europe, που είναι τμήμα του Γενικού Κανονισμού. Υπάρχουν κάποιες ανησυχίες και στα κράτη-μέλη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και η παρούσα πρόταση δεν είναι αποδεκτή. Δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Πάντως η δική μου γνώμη και η δική μου έκκληση μετά από γύρους ολόκληρους διαπραγματεύσεων και συζητήσεων με πολλούς ενδιαφερόμενους είναι ότι η Γενική Διεύθυνση για τις Περιφέρειες και η Γενική Διεύθυνση ΜΟΒ θα πρέπει να καταλήξουν σε κοινή πρόταση που στο μέτρο του δυνατού καλό θα ήταν να διασκεδάσει τις ανησυχίες ώστε να γίνει, δεκτή, να γίνει δεκτός ο γενικός κανονισμός και το στρατηγικό πλαίσιο και να είναι και λειτουργικός. Πάντως, εγώ πιστεύω ότι για να υποστηρίξει πλήρως και το Κοινοβούλιο αυτή την ιδέα θα πρέπει ε, το έγγραφο αυτό να το συνυπογράφουν οι αρμόδιοι επιτροποί Χάν και Κάλλας. Γιατί έτσι θα έχουμε και τα πολιτικά εχέγγυα ότι οι δύο προσεγγίσεις, οι δύο φιλοσοφίες θα υποστηρίζουν, θα στηρίζουν το ΣΥΕΦ. Γιατί ως ε, εισηγητής του Ταμείου Συνοχής μπορώ να δεχτώ τη μεταφορά των 10 δισεκατομμυρίων που είναι τεράστιο κονδύλιο τους άλλους, αλλά θέλω εχέγγυα για τις περιφέρειες, για τα κράτη-μέλη και για την πολιτική συνοχή, αν δεχτώ μια τέτοια μεταφορά. Ευχαριστώ λοιπόν και εκφράζω και πάλι την ευγνωμοσύνη μου προς τους συγκητές για το αξιέπαινο έργο τους. Ο κύριος ε, Λουίς Άλβες. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τους συνεισηγητές για το τιτάνιο έργο τους ε, που ε, ακολουθεί και τη σωστή κατεύθυνση. Ετοιμάζουμε το νέο πλαίσιο προγραμματισμού και το νέο αυτό πλαίσιο είναι πολύ πιο περίπλοκο και στην δομή του και στον ορισμό του αλλά και στην εφαρμογή του. Οι συνεισηγητές πολύ σωστά προσπαθούν από την αρχή να επιτύχουν μια σύγκληση των ε, περιοχών, ώστε στα λειτουργικά προγράμματα που έχουμε εταιρικές συμβάσεις να συμμετέχουν από την αρχή οι περιφέρειες. Θα έχουμε ένα χρόνο περίπου για να προσδιορίσουμε τα λειτουργικά προγράμματα, τα επιχειρησιακά προγράμματα και διανύουμε μια δύσκολη περίοδο ε, και έχουμε και σοβαρή κρίση. Δεν μπορούμε λοιπόν να χάσουμε πολύ χρόνο σε ό,τι αφορά την εκταμείευση των κονδύλιων. Και θα πρέπει πάντως να εμπλέξουμε όλα τα επίπεδα της διακυβέρνησης και το τοπικό και το περιφερειακό στο νέο ε, πλαίσιο προγραμματισμού είναι πολύ σημαντικό για να είναι αποτελεσματικέ οι νέε μα επενδύσεις. Επίσης θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με το θέμα της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουμε ε, στην Ευρώπη που είναι αυτόνομες από οικονομική και διοικητική ε, άποψη για την εκτέλεση των πολιτικών τους και δεν υπάρχουν ανισορροπίες σε αυτή την εφαρμογή. Τώρα να πλήξουμε αυτές τις περιοχές ε, επειδή τα, οι κεντρικές κυβερνήσεις έχουν δημοσιονομικά ελλείμματα ή δεν εφαρμόζουν σωστά τα σύμφωνα σταθερότητας, κατά τη γνώμη μου είναι άδικο και εσφαλμένο. Συμφωνώ λοιπόν με την κατάργηση ε, της μακροοικονομικής αρεσιμότητας και στενίζομαι τη θέση των συνεισηγητών. Τέλος, είναι σημαντικό η πολιτική συνοχής να εξυπηρετεί όντως ε, το στόχο της ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι θεμελιώδης σημασία για όλους. Αλλά χρειαζόμαστε και κάποια ελαστικότητα στην προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή, από τον bottom-up. Γιατί η πολιτική συνοχής εκτός από τους στόχους αυτούς, θα πρέπει να εξυπηρετεί και το στόχο του περιορισμού των ανισοτήτων, της διαφύρωσης των κενών που υπάρχουν μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης, που είναι και η αιτία του κακού σε μεγάλο βαθμό. Γιατί με μια τέτοια ελαστικότητα πιστεύω ότι μπορούμε να ε, μειώσουμε τις ανισότητες μεταξύ των περιφερειών. Και το θέμα των απόμακρων περιοχών και το τι συνέβη με, το τα κονδύλια που έχασαν είναι ένα παράδειγμα που μας δείχνει πόσο θα πρέπει να προσπαθήσουμε για να μειώσουμε αυτές τις ανισότητες που υπάρχουν μεταξύ των περιφερειών. Σας ευχαριστώ. Η Μαριτερέζ Σάντσες Σμιτ. Marie-Thérèse, could somebody just... No, she was not sleeping, ναι. Όχι, ήταν αφηρημένη, δεν ήταν ότι κοιμόταν ε, η Μαρή Τερέζ. Ζητώ συγγνώμη. Να ευχαριστήσω λοιπόν τους εισηγητές για την πρότασή τους που αντικατοπτρίζουν με σωστό τρόπο τις συζητήσεις τις οποίες κάναμε εδώ εδώ και πολλούς μήνες. Χαιρετίζω τις τροποποιήσεις και για τη νομική φάση του κοινού στρατηγικού πλαισίου όπως επίσης και τις προτάσεις για την εξάντερεσιμότητα, για την ε, σύναψη των εταιρικών σχέσεων και ξέρετε ότι με ενδιαφέρουν εμένα ότι έχουν σχέση με τα χωροτακτικά και ε, επίσης προτείνεται η κατάργηση και των καταλόγων των σχετικών με τις αστικές περιοχές και αυτό είναι θετικό. Παρ' όλα αυτά έχω κάποιες απορίες. Μήπως ένα μικρό κομμάτι του άρθρου 21 να το κρατήσουμε έτσι ώστε τα διαρθρωτικά ταμεία να χρησιμοποιούνται και για επενδύσεις που να ευνοούν την ανάπτυξη. 61 ε, με 66 στις τροπολογίες αυτές. Μήπως οι εισηγητές θεωρούν ότι υπάρχει ένας κίνδυνος εξασθένησης του στόχου της θεματολογικής συγκέντρωσης. Σχετικά με το 26 οι εισηγητές προσθέτουν το επίθετο εδαφικός και δεν μπορώ να διαφωνήσω. Γιατί όμως να μην προσθέσουμε όμως την ίδια λέξη, το ίδιο επίθετο και στα λειτουργικά προγράμματα και στις εταιρικές συμβάσεις. Νομίζω ότι η εδαφική διάσταση θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων αυτών. Και περιμένω με πραγματικό ενδιαφέρον τη δεύτερη σειρά των τροπολογιών. Νίλσεν Jans. Thank you very much. Sorry. I will be very brief. I am a new member of the Parliament. Είμαι νέο μέλος του Κοινοβουλίου. Εντυπωσιάζομαι από την εργασία που έχει γίνει μέχρι τώρα, εντυπωσιάζομαι και από το επίπεδο των συζητήσεων και θέλω να ε, συγχαρώ τους συζητητές για αυτά τα οποία προτείνουν σήμερα. Θα ήθελα μόνο λέγοντας ότι είμαι με νέος εδώ, αλλά δεν είμαι νέος στα πλαίσια της εφαρμογής ε, της πολιτικής συνοχής. Το έχω κάνει σαν ε, δήμαρχος και σε άλλα περιφερειακά επίπεδα από τη δεκαετία του 90. Και αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία όταν διαβάζω την πρόταση αυτή και τις τροπολογίες με τις οποίες θα επανέλθουμε είναι η μεγάλη σημασία των περιφερειακών εταιρικών ε, συμβάσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικές για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής. Είναι κρίσιμες για το μέλλον των περιοχών, των περιφερειών, να πετύχουν στην προσπάθεια την οποία κάνουν για την ανάπτυξη. Θα επανέλθω λοιπόν, θα συζητήσουμε τα θέματα των, ε, που προτείνουν οι εισηγητές, αλλά υπογραμμίζω την περιφερειακή διάσταση. Ευχαριστώ. Δεν ήξερα ότι τελικά πάνε αρκετά γρήγορα τα πράγματα. Έχουμε 10 λεπτά στη διάθεσή μας. Δεν ξέρω ε, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να κάνει σχόλια τώρα. Μπορεί να τα κάνει και το απόγευμα, αν θέλει. Thank you very much, uh, Madam. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πρώτα επιθυμώ και εγώ να αποτίσω αληθινό φόρο τιμής στο έργο των εισηγητών. Η πρόταση γενικού κανονισμού ασφαλώς ε, σήμανε σημαντική πρόκληση και λόγω περιπλοκότητας και λόγω ε, μεγέθους. Μακροσκελές κείμενο δηλαδή. Ε, τους τελευταίους δύο μήνες οι εισηγητές μπήκαν στο απαραίτητο βάθος λεπτομέρειας για να μπορέσουν να διατυπώσουν πολύ καλά διατυπωμένες τροπολογίες. Από τη σκοπιά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βέβαια, της Κομισιόν, ε, ορισμένες βέβαια μας απασχολούν, αλλά βλέπουμε όλες ότι αποδίδουν την ε, πλήρη κατανόηση του θέματος από πλευρά των εισηγητών. Και χαιρόμαστε βέβαια και για την στήριξη που δίνεται σε πολλές από τις βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται η πρόταση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κοινών διατάξεων. Από πλευρά τη Κομισιόν είχαμε βέβαια ε, κάπως περιορισμένο χρόνο για να εξετάσουμε όλες τις ε, τροπολογίες οι οποίες ε, αφορούν βέβαια και πολλές υπηρεσίες της Κομισιόν. Γι' αυτό εγώ θα περιοριστώ τώρα στο να σχολιάσω τις ε, πιο σημαντικές από αυτές και εκεί όπου μπορούμε να δώσουμε μια ξεκάθαρη απάντηση. Πρώτα για την αρχή της εταιρική ε, σχέσης και βέβαια χαιρόμαστε για την υποστήριξη που δίνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ενισχύσουμε την αρχή της εταιρικής σχέσης και με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να αναφέρω ότι το προσωπικό της ε, Κομισιόν που εργάζεται επί του κώδικα διοντολογίας έχει ολοκληρώσει τώρα τη ε, διαδικασία έγκρισης στις 24 Απριλίου και το έγγραφο έχει διαβιβαστεί στο Κοινοβούλιο. Άρα πρόκειται για έγγραφο το οποίο περιλαμβάνει το ουσιώδες περιεχόμενο το οποίο θα δώσει στον κώδικα διοντολογίας Code of Conduct η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις ε, ιδέες που θα πρέπει να εφαρμοστούν στην πράξη στις διάφορες ε, προπαρασκευαστικές και εφαρμοστικές φάσεις ε, των προγραμμάτων. Και βέβαια θα θέλαμε πολύ να έχουμε την ευκαιρία να σας υποβάλουμε το σχέδιο αυτό στην Επιτροπή σας σε το χρόνο. Από τις προτινόμενες τροπολογίες φαίνεται να υπάρχει μια πρόθεση ε, να κάνετε μια ε, προσέγγιση δύο επιπέδων στην εταιρική σχέση, κάνοντας μια διαφοροποίηση ανάμεσα στην εμπλοκή περιφερειακών και τοπικών οργάνων και άλλων εταίρων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάποια επιφύλαξη σχετικά με την διατύπωση τουλάχιστον αυτή που προβλέπει τόσο ε, έντονη διαφοροποίηση, διότι έχουμε μια έννοια της ε, partnership που περιλαμβάνει όλους τους ενδιαφερομένους. Και ανάλογα βέβαια με την περιφέρεια θα είναι κάπως διαφορετικά διατυπωμένη αυτή η partnership. Ωστόσο μας ενδιαφέρει να διατηρηθεί αυτή η βασική αρχή της εταιρική σχέσης, αν και βέβαια μπορεί ε, οι διάφοροι φορείς να παίζουν διαφορετικό ρόλο μέσα σε αυτή την εταιρική σχέση. Ένας αριθμός από τις τροπολογίες σας κινούνται προς μια κατεύθυνση που έχει ως στόχο να διευκρινίσει ή να ενισχύσει στοιχεία τα οποία δεχόμαστε. Για την ex ante conditionality, για παράδειγμα, όπου δεχόμαστε την υποστήριξή σας επί της αρχής, θεωρούμε ότι είναι μηχανισμός ο οποίος μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των δαπανών. Είμαστε άλλωστε ανοιχτοί στην πρόταση ενίσχυσης της διασύνδεσης με τον τύπο επενδύσεως νομίζουμε ότι είναι κάτι το οποίο κινείται προς μια κατεύθυνση που ευθυγραμμίζεται και με τον επιδιωκόμενο στόχο. Το ίδιο για το θέμα της relocation του Α61, εκεί όπου δηλαδή γίνεται μέσα στον ε, ε, τομέα του προγραμματισμού. Το ίδιο για την ελεγκτική αρχή που να είναι τμήμα της ίδιας αρχής όπως η Managing Authority το άρθρο 13. Επίσης ε, το πρόσθετο κείμενο εδώ βρίσκουμε ότι συμβαδίζει με τα όσα δέχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα σημαντικό θέμα είναι αυτό της ευκαμψίας, της ε, flexibility στο προγραμματισμό. Εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει πράγματι ανάγκη να υπάρχει πλήρης ευκαμψία υπό ορισμένε περιστάσεις. Κάποιοι άξονες προτεραιότητας που αναφέρονται σε ορισμένες περιφέρειες αυτό μπορεί να βρει σύμφωνη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βλέπουμε ότι σε ορισμένε περιορισμένε περιπτώσει η δυνατότητα χρηματοδότηση χρηματοδοτικών προτεραιοτήτων, δηλαδή από διαφορετικού θεματικού τομεί, μπορεί να έχει μια διαφορά, αλλά αυτό θα πρέπει να περιορίζεται, θα, θα πρέπει να είναι μέσα σε κάποια όρια. Είναι ζήτημα δηλαδή αναλογικότητας, όπου δηλαδή τα όρια της χρηματοδότησης, ή μάλλον η χρηματοδότηση, οι δυνατότητες χρηματοδότησης είναι περιορισμένες ώστε να αποφευθεί ο κίνδυνος υπονόμευσης της λογικής της παρέμβασης και να σχεδιάζονται προγράμματα που να οδηγούν σε ανάπτυξη. Εκεί όπου έχουμε κάποια δυσκολία σε ό,τι αφορά την, τον συνδυασμό είναι η ανάμιξη ταμείων. Για λόγους διαχείρισης τα ταμεία πρέπει να είναι ξεχωριστά και να τηρούνται ξεχωριστά. Και γι' αυτό ο συνδυασμός των ταμείων, των πηγών χρηματοδότησης δηλαδή, οδηγεί σε μια περιπλοκότητα. Ναι, είναι βέβαια δυνατή η διασύνδεση από ταμεία που είναι σε διαφορετικούς άξονες προτεραιότητας, εκεί όπου μπορούν να διασυνδεθούν και βέβαια, όπως θα το έχετε δει, προβλέπουμε στην πρόταση της Κομισιόν τη δυνατότητα ε, μια, ένα επιμέρους εγχείρημα να μπορεί να χρηματοδοτείται από διαφορετικά ταμεία η Κομισιόν θεωρεί ότι δεν υπάρχει ανάγκη μέσα στον ίδιο άξονα προτεραιότητας να γίνεται μια συγχώνευση των πηγών χρηματοδότηση. Τώρα, για τις προτινόμενε τροπολογίες όπου θεωρούμε ότι κάπως σημειώνονται δυσχέρειες. Πρώτα, ο χρόνος παρουσίαση των προγραμμάτων. Προβλέπεται ότι η εταιρική σύμβαση θα αρχίζει να ισχύει μέσα σε ένα εξάμηνο από την έγκριση των κανονισμών και μετά τα επιχειρησιακά προγράμματα θα υποβάλλονται μέσα σε ένα τρίμηνο από την έγκριση της εταιρική σύμβασης. Υπάρχει λοιπόν μια διαδοχική σειρά. Η ένδειξη που έχουμε εδώ είναι ότι η λογική είναι να δοθεί περισσότερη σημασία στην εταιρική σύμβαση ως το βασικό στρατηγικό έγγραφο. Εδώ έχουμε δύο επιφυλάξεις. Αφενός ο χρόνος που θα χρειάζεται. Αν υπάρχει μια διαδοχική σειρά τότε μπαίνει αυτομάτως μέσα στη διαδικασία μια καθυστέρηση στην έγκριση των προγραμμάτων και, έγκριση, και ε, καθυστέρηση επομένω για την έναρξή τους, το startup. Αυτό κατά τη γνώμη της Επιτροπής δεν είναι καλό. Τα προγράμματα πρέπει να εγκρίνονται στο δυνατόν συντομότερα. Δεύτερο, η έννοια ιεράρχηση ανάμεσα στην εταιρική σύμβαση και στο πρόγραμμα. είναι μια πιο περίπλοκη διάρθρωση από το να είναι απλώς η εταιρική σύμβαση και μετά το επιχειρησιακό πρόγραμμα. Αποδίδει άραγε πραγματικά την περιπλοκότητα των, και την ποικιλία των διαφόρων χωρών Μέσα στην πρόταση της Κομισιόν έχουμε βάλει μια ρήτρα για την ανάγκη λήψη υπόψη των διαφορών των ιδιαιτεροτήτων των χωρών μελών. Για παράδειγμα, χώρε μέλη οι οποίε είναι πολύ ομόσπονδε μπορεί τότε να υπάρχει μια άνωθεν προσέγγιση για την εταιρική ε, σύμβαση. Αλλά θα έχει και ένα bottom-up στοιχείο όπου οι περιφέρειες που καθορίζουν τα προγράμματα θα βάζουν αυτά που επιθυμούν μέσα στο πρόγραμμα. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτά δεν ευθυγραμμίζονται με την απαραίτητα λήψη υπόψη αυτής της ποικιλία, αυτή λοιπόν η διαδοχική σειρά των ε, προσεγγίσεων. Και όπως είπα επιφέρει περιττές καθυστερήσεις στην διαδικασία. Είτε λοιπόν κοινή υποβολή ή υποβολή των προγραμμάτων σύντομα μετά από την έγκριση της ειδική Σύμβασης, αυτό επιτρέπει μια συνδυασμένη διαδικασία διαπραγμάτευσης και αποδίδει πολύ περισσότερο αυτό που θέλουμε. Ε, διακόπτη προς. Ε, κύριε Γενική Διευθυντά, με συγχωρείτε. Ας διακόψουμε καλύτερα. Ας διακόψουμε καλύτερα την απάντησή σας και να ε, συνεχίσουμε αμέσως μετά τις ψηφοφορίες το απόγευμα και θα ακούσουμε και τις ε, απαντήσεις των εισηγητών. Θα ήθελα τώρα να περάσω ένα άλλο θέμα. Λυπούμε πολύ που σας διακόπτω. Έχουμε όμως τρεις νομοδοτήσεις σημαντικές για την Επιτροπή Περιφερειακής Αναπτύξεως και που αναφέρονται και στη μελλοντική δημοσιονομική προοπτική. Έχουμε μια μισή ώρα, δηλαδή μισή ώρα για κάθε γνωμοδότηση και αμέσως μετά την παρουσίαση από πλευρά των εισηγητών Όλοι θα θέλουν βέβαια να μιλήσουν. Ε, μπορούμε να αποφασίσουμε λοιπόν πόσο χρόνο θα διαθέσουμε στον καθένα. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλλαγής και Καινοτομίας. Τόμας Πορέμπα. Έχετε το λόγο κύριε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν περάσω στην παρουσίαση της γνωμοδότησής μου, θα ήθελα να πω λίγα εισαγωγικά λόγια για την ε, ιδέα αυτή της συμβολής της δικής μας Επιτροπής στο νομοθετικό πλαίσιο για το 2014-2020. Εκεί η Επιτροπή έχει υποβάλει μια πρόταση κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική πρόοδο, την κοινωνική αλλαγή και την ε, καινοτομία. Ποια είναι η ουσία αυτού του προγράμματος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη συνένωση τριών υπαρχόντων μέσων, του προγράμματος Progress, του προγράμματος Eures και του μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων για την απασχόληση και προτείνει τη συνένωσή τους ε, σε ένα ενιαίο πρόγραμμα σχετικά με την κοινωνική πρόοδο, τι κοινωνικές αλλαγέ και την καινοτομία. Ε, στα πλαίσια της στρατηγικής και του 2020 και την υλοποίηση των στόχων όπως είναι η πρόθεση της γεωγραφικής κινητικότητας, εξυγχρονισμός ε, και αποτελεσματική εφαρμογή της κοινωτικής νομοθεσίας, ε, καλύτερη διαχείριση, ενίσχυση της ευθύνη για την υλοποίηση των στόχων της απασχόλησης, καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και ούτως και το καθεξής. Φυσικά όλοι αυτοί οι στόχοι είναι αξιέπαινοι, αλλά θα μπορούσαμε να προβληματιστούμε για ποια είναι η πραγματική προστιθέμενη αξία αυτής της συνένωσης των τριών μέσων. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήθελε απλώς να διευκολύνει το δικό της έργο, τη δική της διοικητική διαχείριση. Ε, δυστυχώς, κατά τη γνώμη μου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν παρέχει κανένα δεικτικό στοιχείο σχετικά με την προστιθέμενη αξία Τη συνένωση των τριών προγραμμάτων. Επίση, παραλείπει να καταστήσει εμφανή την οριοθέτηση ανάμεσα στι δραστηριότητε που προβλέπονται στο πλαίσιο του νέου προγράμματο και τη στήριξη που παρέχεται μέσω των Ταμείων Συνοχή. Επίση, δεν συμφωνώ γιατί δεν κατανοώ την πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, διεύρυνση του διοικητικού κόστους. Γιατί σε περίοδο λιτότητας και χρηματοπιστωτικής κρίσης πώς να δεχτούμε μία αύξηση του κόστους. Και το νέο ενιαίο πρόγραμμα έχω την αίσθηση ότι θα αυξήσει το κόστος της διαχείρισης. Επίσης, ε, σε ό,τι αφορά την ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για, την, για το δημοσιοποίηση δημοσιονομικό αποθεματικό 5%. Ούτε και εδώ υπάρχουν ε, επαρκείς πληροφορίες και δικαιολόγηση αυτής της πρότασης. Εγώ πρότεινα μια άλλη λύση. Επίσης, ε, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά τα μικροδάνεια ή οι μικροχρηματοδοτήσεις, γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι το 90% των νέων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από αυτή την άποψη η εύκολη πρόσβαση στη μικροχρηματοδότηση είναι ε, τεράστια σημασία για τις ε, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γι' αυτό πρότεινα αυτό το 5% του αποθεματικού να αφιερωθεί στις μικροχρηματοδοτήσεις. Πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη θα συμφωνήσουν με την πρόταση αυτή, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε μόνο 3% για το Progress, το πρόγραμμα Progress, και αντίστοιχα προτείνω για τα πρόγραμματα Εύρες και το πρόγραμμα για τις μικροχρηματοδοτήσεις. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική η πρόταση για τις μικροχρηματοδοτήσεις σε σχέση με την ε, ισχύουσα κατάσταση της χρηματοδότησης. Πιστεύω ότι θα πρέπει να πλουστευτούν όμως και οι διοικητικές διατυπώσεις. Τώρα που έχω κάποιες αφιβολίες. Ε, πιστεύω ότι είναι άκαμπτο το ανώτατο όριο που προτείνεται για τον κοινωνικό πειραματισμό. Το 17% που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Διαθέσιμης Χρηματοδότησης του προγράμματος Progress για την πρόθεση του κοινωνικού προγραμματισμού. Δεν αναφέρει όμως συγκεκριμένους στόχους της κοινωνικής καινοτομίας και του πειραματισμού. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να καταστήσουμε πιο ελαστικό αυτό το άκαμπτο 17% που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να φροντίσει να ε, συγκεντρώσει ποιοτικά στατιστικά στοιχεία και στοιχεία για την αποτελεσματικότητα των διαφόρων προγραμμάτων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το δίκτυο EURES. Νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας και στα προβλήματα των νέων. Ε, και έτσι οι διάφορες δραστηριότητε των προγραμμάτων θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις ιδιαίτερες ε, ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι. Η αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων των προγραμμάτων θα ε, εξασφαλιστεί με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ανάμειξη των περιφερειών από τη φάση της διαμόρφωσης του προγράμματος μέχρι τη φάση της λειτουργίας. Γιατί οι περιφέρειες είναι σημαντικοί παράγοντες και της πολιτικής συνοχής και μπορούν αποτελεσματικά να συμβάλλουν στην δημιουργία καινοτόμων και αποτελεσματικών προγραμμάτων. Θα πρέπει λοιπόν οι περιφέρειες να αναμειχθούν και στα πλαίσια του προγραμματισμού και της κατανομής των κονδυλίων. Επίσης, είναι σημαντική η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού. Είναι πολύ χρήσιμος αυτός ο μηχανισμός της συνεργασίας και στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής. Στη γνωμοδότησή μου, παρόλο που το σκέφτηκα, τελικά δεν ε, επιχείρησα ορισμό της κοινωνικής επιχείρησης. Γιατί δεν μπορούμε να μιλούμε απλώς μόνο για το καταμερισμό των ε, κερδών μεταξύ των ε, μετόχων. Είμαι πάντως ανοιχτός και στη συζήτηση και στις επικοδομητικές παρατηρήσεις κύριε Πρόεδρε και είμαι πεπισμένος ότι θα μπορέσουμε από κοινού να καταρτήσουμε τη γνωμοδότηση, ώστε να αντανακλά τις ε, διάφορες απόψεις ε, με συνεκτικό τρόπο των μελών της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Είναι παρόντες δύο σκιώδεις ηγητέ, ε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλει άλλος κανείς το λόγο για τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση, παρακαλώ να το δηλώσει τώρα. Η ε, κυρία Κάλεμπαχ είναι η πρώτη σκιώδη συγγήτρια για την γνωμοδότηση και παρα... κλείνω εδώ τον κατάλογο των αγορητών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή, του οποίου η γνωμοδότηση περιλαμβάνει πολλά σημαντικά πράγματα που με βρίσκουν σύμφωνοι. Θα έλθω σε λίγε περισσότερες λεπτομέρειες και θα εξηγήσω και σε ποια κατεύθυνση θα κινηθούν οι τροπολογίες δικές μου, δηλαδή των σοσιαλιστών. Συμφωνώ με τον εισηγητή για την συνένωση των ε, κονδυλίων. Όπως τα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι προβληματικό γιατί πρόκειται για τρία διαφορετικά προγράμματα με τρεις διαφορετικούς στόχους και το Συμβούλιο ναι μεν υποσχέθηκε υποστήριξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρόλα αυτά νομίζουμε ότι εμείς πρέπει να ξεκαθαρίσουμε απόλυτα τη θέση μας. Η συνεργασία με τα άλλα ταμεία είναι πολύ στενή. Και για τα προγράμματα Progress, από αυτά ορισμένα μπορούν να γίνουν κοινωνικά προγράμματα. Οι μικροπιστώσεις μπορούν να δίδονται και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Τα τρία προγράμματα δεν πρέπει να επικαλύπτονται ωστόσο, αλλά πρέπει να αποτελούν συμπλήρωση των κυρίων ταμείων. Πιστεύω ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού. Αυτό όμως σημαίνει σαφέστατα διαβούλευση, στενή διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους. Γι' αυτό δεν μου αρέσει η πρότασή σας να αντικατασταθούν οι ε, χώρες μέλη από ε, οργανώσεις. Για το Progress και για τις μη κρατικές οργανώσεις οι οποίες δεν έχουν ομοσπονδίες στο ευρωπαϊκό επίπεδο να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν. Θα κάνουμε λοιπόν σχετική τροπολογία με την έννοια αυτή. Υποστηρίζουμε πλήρως την επιθυμία του εισηγητή να περιλάβει και το τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο στις διαβουλεύσεις θα κάνουμε και εκεί μια συμπλήρωση. Για τον ορισμό της social enterprise θέλουμε να γίνει σαφέστερα η διατύπωση για να μην υπάρξει ο κίνδυνος κάποιες επιχειρήσεις, ίσως επειδή ο ορισμός δεν είναι τόσο ξεκάθαρος, να αποκλείονται. Χαίρομαι που ο εισηγητής αναφέρεται σε ποσοτική και πολιτική και, συγγνώμη, και ποιοτική αξιολόγηση παρελθόντων προγραμμάτων, αν είναι για παράδειγμα μακροπρόθεσμες ή ε, προοπτικές και ούτω καθεξής. Με την έννοια αυτή λοιπόν πρέπει να τονίσουμε ότι δεν πρόκειται μοναχά για την απασχόληση κάθε αυτήν, αλλά κυρίως για υψηλής αξίας απασχόληση. Για τις μικροπιστώσεις, βέβαια η κατανομή μικροπιστώσεων έχει πράγματι σκοπιμότητα για να μπορέσουν να ξαναβρούν δουλειά ορισμένοι. Γεγονός είναι πάντως ότι στην Αυστρία τουλάχιστον έχουν σημειωθεί πολλές αποτυχίες, χρεοκοπίες δηλαδή ε, τέτοιων επιχειρήσεων που ξεκίνησαν με βάση μικροπιστώσεις αυτές και επομένως δημιουργήθηκε μια στρατιά οφειλετών που οφείλουν να επιστρέψουν τα ποσά αυτά. οδηγούνται λοιπόν σε μια ε, ανεργία. Τώρα, για τα ποσοστά. Εσείς ζητείτε μείωση 15%, εμείς θεωρούμε ότι 25% είναι προτιμότερο για τα προγράμματα κοινωνικού πειραματισμού. Για τις εταιρικές σχέσεις, τα χρήματα θα πρέπει να επιστρέφονται, γιατί από αυτά που λαμβάνονται δηλαδή ως μικροπιστώσεις, νομίζουμε ότι το 20% που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σύνολο του συνολικού προϋπολογισμού είναι σωστό ως ε, τάξη μεγέθους. Θέλουμε όσο το δυνατόν λιγότερα χρήματα να δαπανώνται για διοικητικά. Το ποσοστό που αναφέρεται μου φαίνεται σωστό. Η Κομισιόν λέει 3% βέβαια και κάπου θα πρέπει να διαπραγματευτούμε. Για το άρθρο 6 προτείνεται τα πρόσωπα, οι ο όρος πρόσωπα να αντικατασταθεί από τον όρο εργαζόμενοι. Είναι, είναι μόνο σημειολογικό αυτό, γιατί ίσως δημιουργηθεί εντύπωση ότι οι άνθρωποι που ζητούν, αναζητούν απασχόληση και μόλις έχουν τελειώσει την εκπαίδευσή τους, αποκλείονται από αυτά τα προγράμματα κινητικότητα. Προτιμώ λοιπόν να αντικατασταθεί με άλλο τίτλο. Το άλλο τώρα, Ιδίω για του ανηλίκους. Εδώ το ΕΟΡΕΣ αναφέρεται κυρίως στους νεαρούς, ε, στους, ε, στους νέους ενηλίκους. Εκεί πρέπει να διεξαχθούν κάποιες επικοδομητικές συζητήσεις και για την τροπολογία 5. Ο εισηγητής θεωρεί ότι πρέπει να τονιστεί ότι όλα πρέπει να εγκριθούν εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας. Εκεί δεν βλέπω ε, να υπάρχει καμιά αντίρρηση. Ευχαριστώ ήδη από τώρα για την καλή συνεργασία και αναμένω τις προτάσεις σας. Thank you very much. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Καλή Μαντελή. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς λυπάμαι γιατί το σχέδιο της έκθεσης παρουσιάζεται σε αυτή τη φάση γιατί η Επιτροπή, θα έλεγα η βασική στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Επιτροπή Απασχόλησης έχει ήδη προχωρήσει πάρα πολύ στην εξέταση του θέματος. Το θέμα είναι να προχωρήσουμε την ιδέα της διαχείρισης αυτών των εταιρικών προγραμμάτων. Εμείς δεν είμαστε υπέρ της ε, εισαγωγής των υποχρεωτικών ποσοστώσεων για τις διάφορες ε, προτεραιότητες της ΕΡΕΣ. Εμείς θέλουμε να ορίσουμε τις προτεραιότητες αφήνοντας όμως μεγαλύτερη ευελιξία στην κατανομή των πόρων γιατί αλλιώς φοβάμαι ότι θα βρεθούμε με χρήματα τα οποία δεν θα μπορούμε να δαπανίσουμε σε ορισμένους τομείς και χωρίς καθόλου χρήματα σε κάποιους άλλους τομείς. Ενώ αν έχουμε μια ισχυρή εταιρική σχέση τότε θα έχουμε την ασφάλεια θα έλεγα ότι τα χρήματα θα πηγαίνουν εκεί που πρέπει. Έχει επίσης μεγάλη σημασία να διασφαλίσουμε το ότι η καινοτομία και οι πειραματισμοί στον τομέα των κοινωνικών θα στηρίζονται από συγκεκριμένα προγράμματα και όχι από γενικόλογα προγράμματα ευρείας βάσεως. Πρέπει να έχουν μια τοπική πρακτική διάσταση και γι' αυτό ακριβώς ενισχύουμε για μια ακόμη φορά την αρχή αυτή της εταιρικής σχέσης η οποία θα πρέπει να εφαρμόζεται με τον πλέον διαβριμένο τρόπο μη αγνοώντας τους τοπικούς πρωταγωνιστές. Συμμεριζόμεθα την ανησυχία σας για την ε, ενίσχυση των μέσων που είναι διαθέσιμα για την νεότητα που είναι από τα πρώτα θύματα της κρίσης αυτής. Προτείνουμε όπως το έχουμε κάνει με το σύνολο των πολιτικών ομάδων και με την κυρία Στένμπροκ την εισαγωγή ενός τέταρτου πυλώνα στο πρόγραμμα αυτό που να αποφύνεται ειδικά στις πρωτοβουλίες για την νεότητα ε, και να παρουσιάσει μια τέτοια πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό θα πρέπει να περιληφθεί και στη δική μας έκθεση. Τέλος, δεν σας διεφύγει ότι το θέμα της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των διακρίσεων εγκατέλειψαν το πρόγραμμα αυτό και πήγαν στο πρόγραμμα που ασχολείται με την ιδιότητα του πολίτη ή την ηθαγένεια. Εμείς θα θέλαμε τα θέματα αυτά να είναι θα έλεγα εγκάρσιες προτεραιότητες και σε αυτό πάντα το πρόγραμμα. Θα καταθέσουμε τροπολογίες Ελπίζουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μαζί σας όπως το κάνουμε για να καταλήξουμε στις καλύτερες ε, συμβιβαστικές λύσεις και να υπάρξει μια σωστή συνεργασία ανάμεσα στις δύο κοινοβουλευτικές επιτροπές. Πέτ Λούχαν έχει το λόγο, δεν σε είδα προηγουμένως. Είσαι σκιώδης ηγητής. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θεωρώ ότι πρόκειται για κάποιες αλλαγές οι οποίες προτείνονται σε αυτή τη φάση, ριζικές για τον χώρο της εργασίας στην Ευρώπη και για την αγορά εργασίας ιδιαίτερα στα λεγόμενα νέα κράτη-μέλη. Όλοι γνωρίζουμε τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογίας. Ε, κάποιους τομείς εργασιακούς τους περιθωριοποίησε, κάποιους άλλους τους διεύρυνε το βάρος θα έλεγα σε κάποιους ε, τομείς οι οποίοι είναι ιδιαίτερα προχωρημένοι τεχνολογικά ε, έχουν ε, υπάρξει νέες ευκαιρίες που δεν υπήρχαν πριν 10-15 χρόνια. Έχουμε επίσης λοιπόν διαφορετικές ηλικίε ή σειρέ ηλικιών οι οποίες θίγονται από τις αλλαγές αυτές. Είναι απαραίτητο λοιπόν να καταστήσουμε πιο αποτελεσματικές τις περιφερειακές και τις εθνικές πολιτικές οι οποίες έχουν σαν στόχο τα κοινωνικά προβλήματα και πρέπει να υπάρξει και ένας καλύτερος ε, συντονισμός που θα βοηθήσει την ευρυθμότερη λειτουργία της αγοράς εργασίας. Σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να απλοποιήσουμε τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται τα ποσά που είναι στη διάθεσή μας και να καταστήσουμε με τον τρόπο αυτό τα ποσά πιο αποτελεσματικά και να κάνουμε αλλαγές οι οποίες να εξυπηρετούν την καινοτομία και τις αλλαγές όπου αυτές είναι απαραίτητες στον κοινωνικό χώρο. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε και τα τρία υπάρχοντα μέσα να τα αντιμετωπίσουμε ενωτικά. Έουρες, πρόγκρες και τα μέσα, το εργαλείο ή το μέσο μικροχρηματοδότησης. Θα πρέπει λοιπόν ε, να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τα κοινωνικά προβλήματα μέσα από ένα ενιαίο ε, πρόγραμμα το οποίο να λειτουργεί ε, με ολοκληρωμένο τρόπο και όχι με επιμέρους ή αποσπασματικό τρόπο. Τα τρία μέσα λοιπόν που έχουμε στη διάθεσή μας θα πρέπει να τα συντονίσουμε καλύτερα και να βελτιώσουμε τις επιδόσεις τις οποίες έχουμε στον χώρο τον κοινωνικό. Ένας από τους ε, βασικούς στόχους του νέου προγράμματος που προτείνεται είναι ο εξυγχρονισμός της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές ε, ε, ρυθμίσεις οι οποίες έχουν τεθεί σε λειτουργία τον τελευταίο καιρό όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και επιμέρους στις χώρες. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία για τους Ευρωπαίους πολίτες και ιδιαίτερα για τους πολίτες ε, της νοτιοανατολικής Ευρώπης, λέει ο κ. Λούχαν. Ξέρετε ότι οι πολίτες αυτοί δεν μπορούν να αναζητήσουν θέσεις απασχόλησης ε, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια κοινή θέση για τον σωστό συντονισμό των τριών μέσων θα δείτε ότι εδώ θα υπάρξουν διαφορές ανάμεσα στους ευρωβουλευτές, όχι μόνο επί τη βάση της πολιτικής τους ομάδας, αλλά και της εθνικότητάς τους. Οι θέσεις τις οποίες θα καταλήξουν θα εξαρτηθούν από τη χώρα από την οποία προέρχονται. Γι' αυτούς λοιπόν τους λόγους είναι απαραίτητο να υπάρξουν αλλαγές. Γι' αυτούς τους λόγους θα πρέπει οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποστηριχθούν από το μεγαλύτερο ποσοστό Ευρωβουλευτών. Έχουμε τη στρατηγική 2020, έχουμε τη στρατηγική της ολοκληρωμένης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, έχουμε ε, μπροστά μας ε, την εφαρμογή της αρχής της καινοτομίας. Όλα αυτά εφόσον μπορέσουμε να τα προωθήσουμε συνεργαζόμενοι με τα κράτη-μέλη και να τους επιβάλλουμε μια ουσιαστική πολιτική συνοχής και μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης θα χαρακτηρίσει το σύνολο των πολιτικών μας. Αυτά λοιπόν τα καινούργια εν πολλής κοινωνικά μέσα παρέμβασης θα πρέπει να εγγραφούν θα έλεγα στο πεδίο και των υπολείπων τομεακών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που όλες μαζί χαρακτηρίζονται από τους στόχους της στρατηγικής 2020. Να πω λοιπόν ότι η ύπαρξη ενός κανονισμού είναι απόδειξη θα έλεγα αποτελεσματικότητας, αποφασιστικότητας και σωστή στήριξη των κοινωνικών πολιτικών και δείχνουν επίσης την επιθυμία μας να δημιουργήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα σε όλες τις εμπλεκόμενες ομάδες ανεξαρτήτως του επίπεδου από το οποίο προέρχονται ευρωπαϊκό, εθνικό ή περιφερειακό. Στα πλαίσια πάντα επαναλαμβάνω της Ευρώπης 2020, της στρατηγικής 2020. Να υπογραμμίσω επίσης και τη σημασία που έχει η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και η κοινωνική καινοτομία. Εδώ δεν έχουμε μπορέσει να τα πλαισιώσουμε πάρα πολύ καλά και γι' αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ορίσουμε σωστά αυτό που ονομάζουμε κοινωνική καινοτομία. Η πλατφόρμα σαν παράδειγμα για την καταπολέμηση της ένδυας είναι ένα από τα στρατηγικά μέσα για την καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι η καινοτομία μπορεί να είναι ένα βασικό τρόπος για την καταπολέμηση σαν παράδειγμα της γύρανσης του πληθυσμού και φυσικά και άλλων προγραμμάτων ε, στα πλαίσια της καταπολέμησης της φτώχειας, της μείωσης της ανεργίας, ε, νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας ανάλογα με τα νέα στυλ ζωής ε, τα οποία ακολουθούνται σήμερα κτλ. Έχουμε κοινωνικά συστήματα φυσικά ανάμεσα στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους και ίσως θα χρειαστεί να γίνουν ορισμένες προσαρμογές των κανόνων αντίστοιχα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα βοηθήσει όλες τις χώρες. Πάντως, νομίζω το ότι η προσπάθεια συνδυασμού των τριών αυτών μέσων θα δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Αυτό είναι κάτι που θα δείξει, θα φανεί και στις τομεακές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα βοηθήσει επίσης την επίτευξη κατωτέρων αποτελεσμάτων των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να έλθουμε σε ε, στενότερη επαφή από ό,τι το κάνουμε και με τις επαγγελματικές ενώσεις ε, και με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και με τις περιφερειακές αρχές έτσι ώστε να λειτουργήσουμε συνεκτικά σεβόμενοι τις κοινοτικές πολιτικές. Ταυτόχρονα και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και τα όργανα, τα περιφερειακά και τα εθνικά θα πρέπει να είναι επιλέξιμα για προγράμματα κατάρτισης ή επανακατάρτισης και επιμόρφωσης των ενηλίκων. Έτσι θα λάβουμε υπόψη μας τις κοινωνικές αλλαγές. Δεν υπάρχει μια κοινή στάση, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα οικονομικά μέσα, αλλά δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ε, εξειδικεύσεις θα έλεγα για τις διάφορες περιφέρειες ε, ή τις διάφορες χώρες της Ευρώπης, λόγω ακριβώς των συνεπειών ε, της τεχνολογίας και της παγκοσμιοποίησης. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επιτρέψει την καλύτερη προσαρμογή του εργατικού δυναμικού μιας περιφέρειας στις ανάγκες της αγοράς. Στηρίζω λοιπόν τις προτάσεις του εισηγητή. Πιστεύω ότι είναι βέβαια μια περίπλοκη έκθεση, το θέμα είναι περίπλοκο, είναι δύσκολο να καταλήξουμε σε κοινή θέση, είναι απαραίτητο όμως να το πετύχουμε. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά στον κύριο Νίλσεν. Μου αρκεί και ένα λεπτό. Θα ήθελα να τονίσω τη σημασία που έχει ο ορισμός της κοινωνικής επιχείρησης τις προάλλες στην ε, διακομματική ομάδα ε, ε, για την εταιρική ευθύνη είχαμε πολύ μπερδεμένη συζήτηση. Πιστεύω ότι μια κοινωνική επιχείρηση θα πρέπει τα κέρδη της να μην τα μοιράζει στους μετόχους, αλλά να τα επενδύει εκ νέου. Νομίζω ότι είναι αναπόσπαστο στοιχείο της ιδέας μιας κοινωνικής επιχείρησης αυτή η πολιτική. Ευχαριστώ. Ο κύριος Θόμας Πορέμπα, ο εισηγητής μας, παρακαλώ να σχολιάσει αυτά που ακούσαμε. Μπορούμε να ανακεφαλαιώσουμε τη συζήτηση. Ναι, ναι, βέβαια. Ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους ε, για τις παρατηρήσεις ε, που εξέφρασαν ως προς την γνωμοδότησή μου. Θα ήθελα να πω ότι γενικά υποστηρίζω το επίπεδο χρηματοδότηση αυτού του νέου ενιαίου προγράμματος από Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που προτείνει, προκύπτει από τη συνένωση των τριών προηγουμένων. Ε, θα ήθελα πάντως θα πρέπει να αποφύγουμε ε, επικάλυψη με τα περιφερειακά προγράμματα γιατί Πολλέ φορές έχουμε επικάλυψη μεταξύ των δύο πηγών χρηματοδότησης. Θα πρέπει λοιπόν να καταλήξουμε σε μία πρόταση ώστε να αποφύγουμε κάτι τέτοιο, γιατί φυσικά δεν συνάδει με την αποτελεσματικότητα της πρόταση του νέου ενιαίου προγράμματος. Σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό πειραματισμό, από ό,τι γνωρίζω από την προσωπική μου πείρα, δεν καταφέρουν όλες οι χώρες να έχουν πετυχημένο τέτοιο κοινωνικό πειραματισμό και υπάρχει διαφορετικός βαθμός εφαρμογής προγραμμάτων κοινωνικού πειραματισμού. Γι' αυτό και πρότεινα μείωση του ανατάτου ορίου για τέτοιου είδους πειράματα. Αυτό που με ενδιαφέρει κυρίως στη γνωμοδότηση είναι να τονίσω ότι Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να επικεντρωθούμε στους ε, ανθρώπους που ψάχνουν δουλειά, τους νέους, ε, τους ανέργους, ε, που είναι το, το ανθρώπινο δυναμικό και σημαντικό στοιχείο του μέλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι νέοι θα προωθήσουν την κοινωνική ανάπτυξη και την οικονομική ανάπτυξη και αυτούς θα πρέπει να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο. Και πιστεύω ότι τα δικά τους προβλήματα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και αυτό τονίζω στη γνωμοδότησή μου, την ανάγκη να στηρίξουμε τους νέους, κυρίως τους νέους που ψάχνουν δουλειά. Όπως είπα και προηγουμένως, όλες τις παρατηρήσεις που άκουσα θα τις λάβω υπόψη, θα γίνουν συναντήσεις και με τους και οδησηγητές, προκειμένου να διαμορφώσουμε μια συνενετική γνωμοδότηση. Το ζήτημα βέβαια είναι πολύ δύσκολο και συμφωνώ με τον κύριο Πέτρο Λούχαν ότι η αναζήτηση συνενετικής ε, προσέγγισης θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, αλλά δεν είναι και αδύνατο κάτι τέτοιο, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια κοινή βάση, προέκυψε και από τη συζήτηση, πιστεύω ότι, λοιπόν ότι υπάρχουν ελπίδες να καταλήξουμε στη συνενετική γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Ε, thank you ε, very much. Ευχαριστώ πολύ. Μένει να εγκρίνουμε την προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. 3 Μαΐου ας είναι, αυτή προτείνω, 12 το μεσημέρι. Καλά λοιπόν προχωρούμε στο επόμενο θέμα της ε, ημερήσιας διάταξης, την γνωμοδότηση του Ιωακίμ Ζέλερ για το μέσον γειτονία. Μετά από την πρώτη μετά από την πρώτη αυτή παρέμβαση θα ήθελα να σκεφτείτε ποιος άλλος θέλει να λάβει το λόγο. Μετά από τον κύριο Τσέλερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η συνθήκη της ε, ε, λειτουργίας της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει και μια πολιτική γειτονία με 16 χώρες που προτάθηκε και άρχισε να ισχύει εδώ και κάποιο διάστημα. Αίγυπτος, Αρμενία, Αζερβαϊτζάν, Γεωργία, Ισραήλ, Ιορδανία, Λιβύη, Λίβανος, Μαρόκο, Μολδαβία, τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη, Συρία, η Τινησία και η Ουκρανία. Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει στις γειτονικές της χώρες μια προτιμησιακή εταιρική σχέση. με κοινή δέσμευση σε αξίες και αρχές όπως δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα, κράτος δικαίου, χρηστή διακυβέρνηση, αρχές της οικονομίας αγοράς, βιώσιμη ανάπτυξη και δράση για το κλίμα. Η πολιτική αυτή προβλέπει επίσης πολιτική σύνδεση βαθύτερη και βαθύτερη οικονομική ολοκλήρωση, αυξημένη κινητικότητα και βελτίωση διαπροσωπικών επαφών. στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο η πολιτική αυτή θα συνεχιστεί με ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο που θα ισχύσει για όλες τις χώρες εταίρους που θα περιλαμβάνει τώρα και τη Ρωσία. Ήδη στην περίοδο 2007 έως 2013 υπήρξε και για πρώτη φορά κανονισμός σχετικός. Τώρα, η επανεπεξεργασία του νέου αυτού μέσου. Ποιο στόχο έχει. Στα πλαίσια της επανεξέτασης της ε, πολιτικής γειτονίας αναλύθηκαν και αξιολογήθηκαν οι στόχοι. Οι δημόσιες διαβουλεύσεις κατέδειξαν ότι είναι απαραίτητο να γίνουν κάποιες αναπροσαρμογές και αυτές έχουν ληφθεί υπόψη από την Κομισιόν. Και εμείς στην ακρόασή μας για τη διαμεθοριακή συνεργασία Ακούσαμε εμπειρογνώμονες οι οποίοι μας είπαν ότι στο μεταξύ αυτό η διαμεθορική συνεργασία στις παραμεθόριες περιοχές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει σημειώσει επιτυχίες. Ενώ η διαμεθορική συνεργασία στα εξωτερικά όρια της Ένωσης εξακολουθεί να σημειώνει σημαντικές ελλείψεις. Το ίδιο έγιναν ακροάσεις από τον εισηγητή στην Επιτροπή Εξωτερικών, εκεί οι εμειρογνώμονες ε, μας επιβεβαίωσαν ότι η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας χρειάζεται καλύτερο προσανατολισμό για να μπορέσει να επιτύχει τους στόχους της. Τώρα, ποιες είναι οι αναπροσαρμογές οι οποίες πρόκειται να γίνουν. Πρώτα, η εφαρμογή της αρχής more for more. Αυτός είναι ο βασικός πυρήνας των ιδεών που επιτρέπει καλύτερη διαφοροποίηση μεταξύ των χωρών εταίρων, στη βάση δηλαδή της δέσμευσής τους για κοινέ αξίες και προβλέπει οικονομικά ε, κίνητρα για τις χώρες οι οποίες ε, θα κάνουν και τις μεγαλύτερες προσπάθειες. Όχι πλέον ένα απλό πασπάλισμα, μια, μια, ε, ένας κατακαιρματισμός των πόρων, αλλά πιο συγκεντρωμένη πολιτική. Θα μειωθούν οι διάρκειες των προγραμμάτων, θα διασυνδεθούν περισσότερο με τομείς εσωτερικής πολιτικής και περισσότερη διασύνδεση και συνοχή και με τους άλλους μηχανισμούς εξωτερικού εμπορίου. Τώρα, αυτό που έχει σημασία από την πλευρά της περιφερειακής πολιτικής ανάπτυξης, προσπάθησα εγώ να τα περιλάβω στο πλαίσιο και των τροπολογιών που υποβάλλω στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. όπως έδειξε η ακρόαση ή μάλλον όπως έδειξαν οι διαβουλεύσεις είναι απαραίτητο να γίνουν ορισμένες αλλαγές. Μεταξύ αυτών η διεύρυνση του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής για να περιληφθούν ορισμένα σημαντικά πολιτιστικά κέντρα καθώς και η αρχή της κοινή διαχείρισης των πόρων. Άλλες προσαρμογές είναι ωστόσο ακόμη απαραίτητες και τώρα έρχομαι στις τροπολογίες μου. Πρώτα, αύξηση των κονδυλίων για την διαμεθοριακή συνεργασία στο 7% της ε, ε, χρηματοδότησης του ΕΝΗ, του, οργάνου, του εργαλείου δηλαδή για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία. Εδώ υπάρχει και ένα σφάλμα στο σχέδιο της Κομισιόν αναγράφεται ακόμη 3% για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό ε, γειτονία, αλλά δεν ισχύει αυτό το 3%. Είναι ήδη 5% και εμεί είπαμε 7%. Εμεί ζητάμε λοιπόν αύξηση στα 7% των διαθέσιμων πόρων, των διαθέσιμων κονδυλίων και το ζήτησα εγώ. Δεύτερο, αναφορά στην ε, εδαφικότητα και στη συνεργασία στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με, την νέα τροπο, με το νέο τροποποιημένο κανονισμό που μπορούν να χρηματοδοτούνται τώρα εγχειρήματα και στα εξωτερικά σύνορα και να έχουν και διασύνδεση με την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία. Μου φαίνεται εμένα χρήσιμη και απαραίτητη. Η συμπερίληψη του περιφερειακού και τοπικού πλαισίου και της κοινωνίας των πολιτών στα προγράμματα ανάπτυξης, στην βάση δηλαδή εταιρικών συμβάσεων και multi-level governance, ιδίως στο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς επίσης και μη κρατικέ οργανώσεις, ε, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε γειτονικέ χώρες, που θα πρέπει να εμπλέκονται, να συμμετέχουν στον προγραμματισμό και στο σχεδιασμό. Σε πολλές από τις χώρες της γειτονίας βλέπουμε δύσκολες συνθήκες σε ό,τι αφορά τις ε, κεντρικές τους κυβερνήσεις, όμως οι προσπάθειες της πολιτικής της γειτονίας πρέπει να έχουν περισσότερο περιφερειακό χαρακτήρα. Επικρίνω επίσης το κριτήριο του πληθυσμού για την κατανομή των κονδυλίων, όπως αυτό έχει δηλαδή περιληφθεί στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει σε στρέβλωση της κατανομής των κονδυλίων, διότι συχνά περιφέρειες με χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα έχουν ανάγκη το ίδιο από κονδύλια όπως αυτές που έχουν μεγαλύτερη πληθυσμιακή δύναμη. Νομίζω επίσης, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, όπως συνηθίζεται δηλαδή και σε άλλες ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, έτσι και στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία πρέπει να γίνεται μια ενδιάμεση αξιολόγηση, όπως γίνεται και στην πολιτική συνοχή και μάλιστα έχει αποδειχθεί η αξία της πρακτικής αυτής. Και πέρα από αυτό, η κατεξουσιοδότηση πράξης που γνωρίζω ότι επικρίνονται από εμάς συχνά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ωστόσο ε, τις χρησιμοποιεί και είναι εν πάση περιπτώσει καλύτερες από την διατύπωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λέει «in duly justified circumstances». Να γίνεται τότε μόνο η αξιολόγηση, όταν δηλαδή είναι επαρκώς αιτιολογημένες οι περιστάσεις. Αυτό ε, θα επιτρέψει περαιτέρω διακριτική ευχέρεια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που όμως δεν θα μπορεί να ελέγχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μέσω κατεξουσιωτήσεων πράξεων, πράξεων, εκεί δεν θα έχει βέβαια δικαίωμα βέτο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και επίσης και το τονίζω αυτό πάλι, θέλω και το έχω συζητήσει με ορισμένους συναδέλφους της Επιτροπής Εξωτερικών, ζητώ ιδιαίτερο κανονισμό για την διαμεθοριακή συνεργασία. Στην τροπολογία 1 το περιλαμβάνω αυτό. Για την διαμεθοριακή συνεργασία με τις χώρες της γειτονίας, αυτή είναι πολύ περιορισμένη και συχνά χαμηλής ποιότητας. Γι' αυτό χρειάζεται ένας ξεκάθαρος ορισμός για το τι σημαίνει κοινό έργο, καθώς επίσης και τι σημαίνει κοινή χρηματοδότηση. Εκεί θα χρειαστεί ένα κοινό λογαριασμός, καθώς και κοινά κριτήρια της επιλεξιμότητας. Αυτά μπορεί να γίνουν σε κανονισμό ή μπορεί να γίνουν σε ιδιαίτερο κανονισμό για την διαμεθοριακή συνεργασία μέσα στα πλαίσια της πολιτικής συνοχή. Το ίδιο εδώ όπω και για την πολιτική γειτονία αρχικά προβλεπόταν ιδιαίτερο κεφάλαιο. Αλλά τώρα προτείνεται ιδιαίτερος κανονισμός και αυτό μπορεί να ισχύσει και για το εργαλείο γειτονία. Για να βελτιωθεί η συνεργασία επαναλαμβάνω ότι είναι χρήσιμο και επιθυμητό να υπάρξει ε, ξεχωριστός κανονισμός. Αυτά σαν μια πρώτη προκατακτική τοποθέτηση. Το έγγραφο εργασίας για το εργαλείο γειτονίας Ακόμα δεν το έχει λάβει η Επιτροπή Εξωτερικών. Όμως είμαι σε επαφή με τον εισηγητή τους, κύριο Μπούκαν, και με τους κοιόδης εισηγητές εδώ στη δική μας Επιτροπή, όπου έκανα χθε μια πρώτη συνάντηση και μια πρώτη διαβούλευση. Και αναμένω βεβαίως τις παραπέρα συζητήσεις. Uh, Ευχαριστώ. Έχουμε παρόντες δύο ε, σκιώδεις ηγητές. Δεν ξέρω αν θέλει κανείς άλλος να λάβει μέρος στη συζήτηση για να κλείσει ο κατάλογος παρακαλώ. Και ένας ομίλητης πέραν των σκιωδών εισηγητών. Ο Ευγέννη Κυρίλοφ είναι ο πρώτος σκιώδης εισηγητής. Uh, Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Σέλερ για την uh, εισαγωγή του Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω αυτό το οποίο ζήτησε για περισσότερη διασυνοριακή συνεργασία. Η συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη ή ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τρίτες χώρες είναι χαρακτηριστικό θα έλεγα σημείο πολιτικής συνεργασίας, οικονομικής συνεργασίας, αναπτυξιακής συνεργασίας και ταυτόχρονα δημιουργεί ευκαιρίες για την εφαρμογή περισσότερων προγραμμάτων και οδηγεί σε καλύτερες σχέσεις ανάμεσα στις χώρες αυτές και μερικές φορές όταν υπάρχουν ακόμα και κάποιες συγκρούσεις συνεισφέρει στην οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης και στην αποκατάσταση των επαφών ανάμεσα στους λαούς κάτι το οποίο έχει μεγάλη σημασία. Συζητήσαμε λοιπόν χθες με τον κύριο Ζέλερ και την πρότασή του. Καταλήξαμε σε αρκετές συμφωνίες. Έχουμε ελάχιστε διαφορές τις οποίες θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε με κάποιες από τις τροπολογίες αλλά αυτό το οποίο απαιτείται είναι σωστότερη ισορροπία. Το θέμα είναι να μην ζητάμε από τις γειτονικές χώρες περισσότερα από όσα μπορούν να προσφέρουν. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τις διαφορές οι οποίες υπάρχουν. Καταρχάς, με διαφορετικό τρόπο βλέπει τις ε, γειτονικές σχέσεις κανείς με τους ανατολικούς ε, εταίρους, αλλά με διαφορετικό τρόπο βλέπει τις σχέσεις μας με τις γειτονικές χώρες, σαν παράδειγμα της Βορειοαφρικής. Αν δούμε ποιες είναι οι ομοιότητες στο μηχανισμό εφαρμογής ε, στα πλαίσια των μέσων συνοχής και στα πλαίσια του μέσου αυτού γειτονίας, θα πρέπει να μην αγνοούμε παράλληλα τα διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης αυτών των χωρών, κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα σε ορισμένες περιπτώσεις και μπορεί να οδηγεί και σε πάρα πολλές μορφές δυσθυμίας της εφαρμογής των μεμονωμένων προγραμμάτων. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν η εφαρμογή της αρχής της εταιρικότητας και στα πλαίσια της εφαρμογής των προγραμμάτων και στα πλαίσια της παρακολούθησης της εφαρμογής των προγραμμάτων δημιουργεί κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πιο αντικειμενικοί. Ένα πράγμα είναι να βλέπει κανείς τις ΜΚΙΟ να συμμετέχουν σε προσπάθειες στη Γεωργία, στην Μολδαβία κτλ. Και εντελώς διαφορετικό να προχωρούμε σε τέτοιου είδους ε, προχωρημένες εταιρικέ συμβάσεις με τη Λιβύη, όπου τα πράγματα εκεί είναι εντελώς διαφορετικά. Κάτι τέτοιο βοηθά σίγουρα τις χώρες αυτές, αλλά σίγουρα δημιουργεί μια κάποια δισκαμψία στις σχέσεις μας με αυτές τις χώρες. Συμφωνώ λοιπόν για την σημασία που έχει η εφαρμογή αυτής της αρχής Ταυτόχρονα όμως δεν θα πρέπει να αγνοούμε κάποια από τα όρια τα οποία υπάρχουν Ίσως θα πρέπει να δούμε εδώ κάποιες τροπολογίες πιθανώς για να καλύψουμε τα κενά. και θα πρέπει η αρχή του περισσότερο για περισσότερα, το more for more, ανάλογα με τις ανάγκες των διαφόρων χωρών, να ισχύσει σε όλες τις περιπτώσεις. Ίσως να υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις οι οποίες ε, πράγματι να μην ε, δέχονται αυτή την αρχή αν θέλετε. Ίσως κάπου ε, το less for less να είναι και χρήσιμο, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις το more for more είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο. Δεν θα είναι εύκολη εν πάση περιπτώσει η διαδικασία αυτής της συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες και μέσα από το καινούριο αυτό εργαλείο γιατί συμπεριλαμβάνει και εταίρους εξοκυβερνητικούς. Απ' την άλλη δεν μπορούμε εμείς να περιοριστούμε στις δυνατότητες που έχουν οι βασικές συγκεντρωτικές αρχές αυτών των χωρών. Πρόκειται λοιπόν για ένα έγγραφο σημαντικό πολιτικά και στην οικονομική του διάσταση το κείμενο αυτό έχει μεγάλη σημασία και ελπίζω να οδηγήσει σε παραγωγικές για όλους και χρήσιμες συμφωνίες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Αλφόνση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω φυσικά τον εισηγητή τον κύριο Τζέλερ για το έργο του. Νομίζω ότι σωστά εντόπισε τα ουσιώδη στοιχεία προκειμένου να βελτιωθεί η πολιτική γειτονία για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού και όλες οι προτάσεις που λέει για την ανάδειξη του ρόλου των περιοχών, για την πολυπίπεδη κυβέρνηση, για τη θέση της κοινωνίας των πολιτών, με βρίσκουν σύμφωνο. Δεν συμφωνώ με τον κύριο Κυρίλοφ. Μην ξεχνάτε ότι αυτός ο προγραμματισμός ε, φτάνει μέχρι το 2020 και ευελπιστούμε ότι μέχρι το 2020 θα έχουν σημειώσει πρόοδο όλε οι, οι χώρες της γειτονίας ό,τι αφορά την κοινωνία των πολιτών και τη δημοκρατία. Οπότε στόχο μα είναι να θεσπίσουμε μηχανισμού για να ενθαρρύνουμε τέτοια σχέδια και να δώσουμε άμεσε προοπτικές μέσω τη συνεργασία τη χώρες τη πολιτική γειτονία. Φυσικά συμφωνώ και με την πρόταση του κυρίου Τζέλερ για τον μη αποκλειστικό χαρακτήρα του, κριτήριου, του πληθυσμιακού κριτηρίου δεν θα πρέπει να περιοριζόμαστε μόνο σε αυτό το πληθυσμιακό κριτήριο, γιατί έχουμε μεγάλες περιφέρειες ε, αεροκατοικημένε όμω και το θέμα της χωροταξίας και η πολιτική μεταφορών είναι σημαντικές και δεν θα πρέπει να περιοριζόμαστε μόνο στο πληθυσμιακό κριτήριο, θα μας οδηγήσει σε λάθος αποτελέσματα. Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες και πώς ε, θα συνεργαστούμε με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για την πολιτική γειτονία. Νομίζω ότι η συνεργασία αυτή περνάει μέσα από τη μακροπεριφερειακή στρατηγική. Θέλουμε κάποιε διευκρινήσει λοιπόν που λείπουν προ το παρόν και κάποιε φιλοδοξίε ό,τι αφορά τη μακροπεριφερειακή στρατηγική για να εξασφαλίσουμε συνεργασία, συνέργεια μεταξύ του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, ε, του, Κοινωνικού, του Ταμείου Συνοχής και του μηχανισμού αυτού για την ε, πολιτική γειτονία. Ο κύριος Γιώσεφ Ματού. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η πρόταση κανονισμού στηρίζεται σε μια νέα στρατηγική για την πολιτική γειτονία. Μια στρατηγική που προσαρμόζεται στο νέο πολιτικό πλαίσιο αλλά και στους ε, στόχους, τους ειδικούς στόχους που περιορίστηκαν από 29 στους 6. Ε, εδώ δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην αρχή more for more, περισσότερα για περισσότερα, γιατί με την αρχή αυτή θα γίνει καλύτερη διαφοροποίηση μεταξύ των χωρών εταίρων και των σχέσεών τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί εδώ επιβραβεύεται η αξία. Θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφο Τσέλερ γιατί κατάφερε να συμπεριλάβει στη γραμμάτωσή του όλα τα βασικά στοιχεία του μελλοντικού κανονισμού. Ένα μικρό πρόβλημα υπάρχει μόνο που πιστεύω ότι θα διαθετηθεί στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Καλό είναι όμως να το επισημαίνουμε και εμείς. Σε ό,τι αφορά αυτό το μηχανισμό της ε, γειτονίας, τι θα γίνει αν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσει να κόψει τις πολιτικές γέφυρες με ορισμένα καθεστώτα. Είμαι ο συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού για το θέμα αυτό και πιστεύω ότι σε τέτοια περίπτωση καλό θα ήταν να συνεχιστούν οι διαπροσωπικές σχέσεις και να συνεχιστούν και τα διασυνοριακά προγράμματα. καλό θα ήταν να κρατήσουμε τους δεσμούς μας με την κοινωνία των πολιτών και με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις των χωρών αυτών. Και το λέω αυτό γιατί κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα είδος πολιτιστικής διπλωματίας και να προωθήσουμε τις κοινοτικέ ενωσιακές μας αξίες παρόλο που μερικά πολιτικά καθεστώτα μας δημιουργούν προβλήματα. Γιατί ε, τα πολιτικά προβλήματα έρχονται και παρέρχονται, αλλά οι πολίτες μένουν. Αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνούμε. Ε, γι' αυτό θα υποβάλω και τροπολογία για τον πολιτισμό και την ε, παιδεία. Η, η πολιτιστική συνεργασία και η συνεργασία σε εκπαιδευτικά θέματα είναι σημαντική ειδική στόχη και θα πρέπει να συμπεριληφθούν στα περιφερειακά προγράμματα. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια στον εισηγητή μας. Thank you very much. Ευχαριστώ κύριο Τσέλερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους παρεμβάντες καθώς και τους κυριοδησίγητες. Θα συνδέσω τα όσα είπαν οι κύριοι Κυριλόφ και Ματούλα. Ακριβώς επειδή δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ποιες θα είναι οι πολιτικές εξελίξεις στις διάφορες χώρες, για αυτό το λόγο θεωρώ ότι το εργαλείο της γειτονία πρέπει να μπορεί να εφαρμόζεται με τρόπο διαφοροποιημένο. Και γι' αυτό κάνω και τις προτάσεις που κάνω, δηλαδή να προσανατολιστεί σε περισσότερα επίπεδα στρατηγικές δηλαδή περισσότερων επιπέδων, multi-level governance, μη κρατικέ οργανώσεις κλπ. Με μια χώρα de facto οι πολιτικές σχέσεις έχουν διακοπεί, με τη Λευκορωσία δηλαδή. Όμως η μοίρα των πολιτών, των ανθρώπων στη Λευκορωσία δεν μπορεί να μας αφήσει αδιάφορους. Πρέπει λοιπόν να μπορούμε να αντιδράσουμε με τρόπο εύκαμπτο. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε και μια ερμηνεία του εργαλείου της ε, γειτονίας που να αποσυνδεθεί από το τι κάνουν οι κεντρικές κυβερνήσεις. Θυμίζω και μια συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο προέτους περίπου όταν είχε αρχίσει η λεγόμενη Αραβική Άνοιξη. Πολλοί ήταν τότε εκείνοι που είπαν μέσα σε μεγάλη εφορία ότι πρέπει να ενισχυθούν οι χρηματοδοτήσεις που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ορισμένες αραβικές χώρες. Είχαν πει τότε ορισμένοι μάλιστα να πάρουμε και κονδύλια από την ανατολική γειτονία και να τα διοχετεύσουμε στις χώρες της Μεσογείου. Όμως οι εξελίξεις που ακολούθησαν μετά μάλλον δείχνουν ότι αυτά όλα θα ήταν περιτά και μάταια. Αν είχαμε δηλαδή λάβει υπόψη μόνο τις εξελίξεις εκείνες. Χρειάζεται λοιπόν μια εμβάθυνση ε, τη συζήτηση και μια συζήτηση που πρέπει να γίνει και με την Επιτροπή Εξωτερικών. Εμείς άλλωστε δίνουμε μόνο εντό εισαγωγικών γνωμοδότηση από την περιφερειακή, ε, από τη σκοπιά μάλλον τη περιφερειακή ανάπτυξη. Βεβαίω είναι πολύ σημαντική αυτή. Η σύνδεση τώρα Ρέγκι και Άφετ είπα ότι την κάνω εγώ τη διασύνδεση αυτή γιατί συναντώμαι με τον εισηγητή του και θα συνδεθώ όλο και συχνότερα το επόμενο διάστημα. Ακόμα δεν έχουν δημοσιεύσει το δικό τους έγγραφο. Εάν τώρα μπορέσουμε να δράσουμε και να αντιδράσουμε γρήγορα, μπορεί να περιληφθεί η γνωμοδότησή μας και στο έγγραφο που θα ετοιμάσει η ε, Επιτροπή ΑΦΕΤ. Ο κ. Αλφονσίν μίλησε για τις μακροοικονομικές στρατηγικές. Και εγώ ε, διαρωτήθηκα κατά πόσο θα τις βάλουμε μέσα. Το ζήτημα είναι τώρα το εξή ότι έχουμε μια μακροοικονομική στρατηγική εγκεκριμένη, που είναι αυτή της Βαλτικής γίνεται στην ουσία μόνο μεταξύ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μια εξαίρεση τη Ρωσία όπου ήδη εκεί αναπτύσσονται κάποιες ιδέες για την εδαφική συνεργασία που σύμφωνα με τις απόψεις των εμπειρογνωμόνων πάντως μέχρι τώρα δεν έχει αποβεί επιτυχής. Άρα υπάρχει σημαντική ανάγκη βελτίωσης και παρόλο που έχουν δοθεί σημαντικά κονδύλια. Τώρα κατά πόσον αυτό μπορεί να συνδεθεί με τη μακροοικονομική αυτή στρατηγική με την συγγνώμη, μακροπεριφερειακή στρατηγική, ε, αυτό ακόμα δεν είναι γνωστό. Υπάρχουν κάποιες προσεγγίσεις μακροπεριφερειακής συνεργασίας και για τις πολιτικές των χωρών γειτονία. Έχουμε τη μακροπεριφερειακή συνεργασία του χώρου του Δούναβη με συμμετοχή χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βαλκανικής Χερσονήσου που δεν εμπλέκονται όμως σε πολιτική γειτονία, αλλά σε αυτά που συζητούμε τώρα, δηλαδή στη στατηγική της ένταξης. Πρόκειται για άλλη στατηγική προσέγγιση που τα σχετικά τα λέει η κυρία Λουκατσιεύσκα. Και η άλλη μακροπεριφερειακή στρατηγική είναι η Ατλαντική. Πάλι με χώρες που εντάσσονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα εδώ εγώ τα έχω αφήσει αυτά απ' έξω από την έκθεσή μου, διότι δεν βλέπω σχέδια μακροπεριφερειακής στρατηγικής να μπορούν να εφαρμοστούν σε χώρες που συμμετέχουν στην πολιτική γειτονία. Σας ευχαριστώ κατά τα άλλα, ευχαριστώ και τους ε, συμβούλους και όλους όσοι συνέβαλαν στην σύνταξη της έκθεσής μου. μέσα από μια πολύ ευρία διαδικασία διαβούλευσης. Ευχαριστώ και τους συνεργάτες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικών Δράσεων καθώς και τους αξιωματούχους της Κομισιόν οι οποίοι ε, με τη συμβολή τους μου επέτρεψαν να καταλήξω στο ε, σχέδιο που σας υπέβαλα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα πρέπει να αποφασίσουμε την προθεσμία για τις τροπολογίες, αλλά προηγουμένως να υποβάλω κι εγώ ένα σχόλιο. Στις τροπολογίες, καλό θα ήταν να λάβουμε υπόψη που οφείλεται η αναποτελεσματικότητα των ε, υφιστάμενων προγραμμάτων. Ιδιαίτερα σε ό,τι φορά τα κονδύλια του Περιφερειακού Ταμείου. Είναι σημαντικό να παρακολουθούμε πώς αξιοποιούνται τα κονδύλια. 27 Απριλίου το μεσημέρι, 12 το μεσημέρι λίγη η προθεσμία για τις τροπολογίες. 27 Απριλίου 12 το μεσημέρι και περνάμε στην τελευταία γνωμοδότηση για το πρωί. Μαρή Τερέ, συγγνώμη, τι θέλες. Αύριο είναι 27. Σωστά, αύριο είναι. Εκτός μικροφώνου δυστυχώς τα σχόλια της κυρία Σμιτ. Ναι. Το έλεξα και με τη γραμματεία. Θέλουμε περισσότερο χρόνο για την ε, αναζήτηση συμβιβαστικών προτάσεων. Αύριο Παρασκευή, 12 το μεσημέρι. Να μην χάσουμε όμως την επόμενη εβδομάδα. Αυτό φοβάμαι αν παρατείνουμε την ε, ε, προθεσμία για τις τροπολογίες, γιατί την επόμενη εβδομάδα θα αποσιάζουμε. Δεν ξέρω, η γραμματεία... 3 Μαΐου το πολύ, αν θέλετε, παράταση. Οι σκιώδες ηγητές προτείνουν να λήξει αύριο η προθεσμία. Αν όμως προτιμάτε την 3η Μαΐου, η διαφορά είναι ελάχιστη. Ναι, απλώς ε, θέλουν οι σκιώδες ηγητές περισσότερο χρόνο για να μπορέσουν να καταλήξουν σε συμβαστικές ανθρωπολογίες και συμβαστικές προτάσεις. Δεν ξέρω. Αύριο ή 3 Μαΐου. Έτσι όμως περιορίζουμε το χρόνο των σχεδόν εισηγητών να βρουν συμβαστικές τροπολογίες. Εγώ περιμένω από σα ε, συστάσει. Τι προτείνουν οι σκιώδε συγκεκριτές. Εντάξει, 3 Μαου. Ωραία, ευχαριστούμε Μαρή Τερές. Μαριτερέ. 3η Μαΐου λοιπόν ε, η προθεσμία για τις τροπολογίες. Περνάμε στην γραμματότητα της κυρίας Γουκατσιεύσκα για το μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας. Έχετε το λόγο κυρία Γουκατσιεύσκα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ένα σχέδιο κανονισμού με το νομοθετικό πλαίσιο για το νέο μηχανισμό προταξιακής βοήθειας στα πλαίσια των νέων δημοσιονομικών προοπτικών του 2014-2020. Ο μηχανισμός αυτός αφορά τις υποψήφιες χώρες και τις δυνάμει υποψήφιες χώρες για ένταξη. Η Αλβανία δηλαδή, η Βοσνία η Ισλανδία, Κωσυφοπαίδιο, Μαυροβούνιο, Σερβία, Τουρκία, καθώς και η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η γνωμοδότησή μου στηρίζεται σε εκτενείς διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους ε, προσώπους των Γενικών Διευθύνσεων Διεύρυνσης και Περιφερειακής Ανάπτυξης, με ε, αντιπροσωπείς Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σερβία, στην Ισλανδία και αποστολές των υποψηφίων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης ζήτησα τη γνώμη και πολλών κυβερνητικών οργανώσεων από την Αλβανία, τη Μακεδονία, την Τουρκία και το Μαυροβούνιο. Συναντήθηκα και με τον ε, κύριο εισηγητή, τον κύριο ε, Βιγγένιν από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και είχα και συναντήσει με του σκιώδει ηγητέ τη δική μα Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξη. Η γνωμοδότησή μου επίση ε, είναι καρπό ε, συνεργασία και με τον ε, κύριο Τσέλερ γιατί σε πολλές περιπτώσεις και οι δύο γνωμοδοτήσεις είναι συμπληρωματικές. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τη συνεργασία, να ευχαριστήσω και τους συνεργάτε μου και τη γραμματεία της Επιτροπής για την ε, βοήθειά της. Ε, να ευχαριστήσω επίσης και τους συμβούλους μας. Ο μηχανισμός προνταξιακής βοήθειας προσφέρει ε, συνδρομή στις υποψήφιες για ένταξη χώρες. Στόχο έχει την σταθερότητα, την προστασία και την κοινωνική και οικονομική ευμάρεια στις υποψήφιες για ένταξη χώρες ή τις δυνάμει υποψήφιες χώρες, προκειμένου να ετοιμαστούν για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η βοήθεια αυτή θα πρέπει να είναι στρατηγική, αποτελεσματική και στοχευμένη. Ο νέο μηχανισμό προδεξιακή βοήθεια θα πρέπει να λειτουργεί ελαστικά και να λαμβάνει υπόψη τι ιδιαιτερότητε τη κάθε υποψηφία χώρα ή δυνάμει υποψηφία χώρα. Πιστεύω ακράδαντα πάντω ότι είναι σημαντική η ανάγκη για συνέχιση της παροχής τεχνικής και χρηματοδοτικής συνδρομής των υποψηφίων για ένταξη χωρών, γιατί η συνδρομή αυτή συμβάλλει στην ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της πολιτικής εξωτερικών υποθέσεων και διεύρυνσης και συμβάλλει στη σταθερότητα στις γειτονικέ χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρόκειται να σχολιάσω αναλυτικά τις 13 τροπολογίες. Ε, μπορείτε να διαβάσετε στο έγγραφο εργασία και την αιτιολόγηση της κάθε τροπολογίας. Εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ στις ε, τρεις βασικότερες πτυχές της γνωμοδότησής μου. Το πρώτο σημείο αφορά την διασυνοριακή συνεργασία. Η διασυνοριακή συνεργασία αναφέρεται πολύ συχνά στη συζητήση της Επιτροπής μας. Είναι ανεκτήμητο μέσο για την πρόθεση της συνεργασίας μεταξύ των περιφερειών και με το, τη συνεργασία των χωρών με την ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων και των πρακτικών. Η διασυνοριακή συνεργασία μπορεί να αποτελέσει ένα λόγο προαγωγής ε, της ανάπτυξης των πιο μειονεκτικών περιοχών, εξασφαλίζοντας πρόσβασή τους σε τεχνογνωσία και σε πληροφορίες ε, που κατέχουν πιο ανεπτυγμένες περιοχές των κρατών μελών. Από αυτή την άποψη, η γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επικεντρώνεται σε ένα νευραλγικό στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είναι η διεύρυνση. Γι' αυτό και θα πρέπει να εφοδιαστεί η υλοποίηση αυτού του στόχου με πολύ περισσότερα κονδύλια. Όπως και ο κύριο Τσέλερ και εγώ πρότεινα αντί για 3% 7% του ποσοστού αναφοράς για τη διασυνοριακή συνεργασία. Ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο της γνωμοδότησής μου αφορά τα κριτήρια για την κατανομή κονδυλίων από το Μηχανισμό Προδεξιακής Βοήθειας. Κατά τη γνώμη μου, η παρούσα πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, δεν λαμβάνει υπόψη πολύ σημαντικά κριτήρια και πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνεται μια καλύτερη διευκρίνηση και συγκεκριμενοποίηση των κριτηρίων γιατί είναι κάπως πιο γενικά. Ε, φυσικά έχουμε και τον ε, κανονισμό για την ε, εδαφική συνεργασία, βασικό κριτήριο εκείνο το πληθυσμιακό κριτήριο, ενώ σε άλλα σημεία του κανονισμού υπάρχουν προτάσεις το ύψος των κονδυλίων που λαμβάνει μια χώρα να εξαρτάται από, από τη δυνατότητα απορρόφησης και διοικητικής ικανότητας των χωρών. Και στι δύο περιπτώσεις θεωρώ ότι αυτά τα δύο κριτήρια καλό θα ήταν να συγκεκριμενοποιηθούν περαιτέρω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να λάβουν υπόψη και τις ιδιαιτερότητες ή τις ιδιαίτερες ανάγκες ε, των διαφόρων χωρών. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων ε, που πολύ πρόσφατα ε, ξεπέρασαν τον πόλεμο μετά τη διάσπαση της Ιουκοσλαβίας και έχουν πολύ χειρότερες ε, διοικητικές ικανότητες ε, και δυναμικό με άλλες χώρες που είναι πολύ πιο προχωρημένες. Επίσης δεν μπορούμε να λαμβάνουμε το πληθυσμιακό κριτήριο γιατί έχουμε πικροκατοικημένες χώρες όπως η Τουρκία και αεροκατοικημένες όπως η Ισλανδία. Άλλο σημαντικό θέμα της γνωμοδότησης είναι ο ρόλος, ο σημαντικός ρόλος της κοινωνίας των πολιτών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων στις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες. Θα ήθελα αυτές οι οργανώσεις των πολιτών να τύχουν ιδιαίτερης υποστήριξης από το Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας, ώστε να ενισχυθεί και η ικανότητα απορρόφησης, αλλά και η διοικητική ικανότητα των χώρων αυτών και να διαμορφωθεί μια πραγματικά δημοκρατική κοινωνία στις χώρες αυτές. Αυτά λοιπόν είναι τα κύρια σημεία της γνωμοδότησης. Φυσικά θα βρείτε και κάποιες αναφορές για την, για την προστασία των μειονοτήτων, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά και τους μηχανισμούς ε, εμπέδωσης της δημοκρατίας. Ευχαριστώ και πάλι στενά, ε, ευχαριστώ θερμά τους ε, συνεργάτες για τη στενή συνεργασία και τους συναδέλφους και είμαι πρόθυμη να ακούσω τις προτάσεις σας και τα σχόλιά σας με ανυπομονησία. Τρεις εγγεγραμμένοι. Κανεί uh, uh, Κανείς άλλος? Λάβετε υπόψη το γεγονός ότι είσαστε τρεις και έχουμε 25 λεπτά. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για τη θαυμάσια εκθεσή της όπου αναφέρεται σε ορισμένα σημαντικά θέματα για παράδειγμα πάλι τη σημασία των διαμεθοριακών συνεργασιών, κοινά έργα δηλαδή, που μας ενδιαφέρουν εμάς πολύ, με κοινή τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη. Άλλο σημαντικό για μένα είναι το θέμα της δημοκρατίας και ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ιδιαίτερα για ορισμένες από τις χώρες που οδεύουν προς την ένταξη, χώρες διεύρυνση δηλαδή, κυρίως των Δυτικών Βαλκανίων, αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Το άλλο, για πολλές χώρες που βρίσκονται στη φάση της προένταξης, είναι η υποδομή, μάλλον η έλλειψή τη, όπου μένουν πολλά πράγματα να γίνουν, για παράδειγμα για τι επικοινωνίε. Συστήματα επικοινωνιών, επίσης ε, διασυνδέσει ευρέω φάσματο. Εκεί μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο η Ένωση. Το άλλο είναι τώρα η λεγόμενη capacity building για τις κυβερνητικές υπηρεσίες αλλά και για τις μη κρατικές οργανώσεις. Ορισμένες από τις χώρες της προένταξης ακόμα δεν είναι αρκετά ανεπτυγμένες και εκεί χρειάζονται ενίσχυση. Τέλος, που νομίζω ένα θέμα τέτοιο δεν έχει περιληφθεί επαρκώς, για εγκληματικότητα και διαφθορά εξακολουθεί σε ορισμένε από τι χώρε αυτέ να είναι μέγα θέμα. Πρέπει να εξεταστούν λοιπόν και τα νομικά συστήματα και οι πολιτικέ κρατικών προμηθειών, για παράδειγμα, και εκεί πάλι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο να βοηθήσει τι χώρε αυτέ να βελτιώσουν τα συστήματά του, όπω είπα, των δημοσίων προμηθειών, τη καταπολέμηση τη διαφθορά, τη καταπολέμηση τη εγκληματικότητα. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία πρέπει να υποστηριχθούν. Ούτζιας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αντικαθιστώ τον κύριο Γιώβινε ο οποίος είναι απασχολημένος. Οι φιλελεύθεροι και ο Γιώβινε συμφωνούν εν με τις θέσεις τις οποίες παρουσίασε η συγγήτρια Προσυπογράφουμε λοιπόν και τα θέματα τα οποία έχουν τεθεί και την κριτική η οποία ασκήθηκε σχετικά με την προώθηση της διαμεθοριακής συνεργασίας, την ενίσχυση της δημοκρατίας, τον σεβασμό της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θα πρέπει να είναι συμβατές με το τι ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως επίσης και η σωστή κατανομή των κριτηρίων που θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένοι στις τοπικές ανάγκες έτσι ώστε να μην δημιουργούνται μειονεκτήματα ή μειονεκτικές θέσεις σε οποιαδήποτε χώρα ιδιαίτερα αν είναι υποψήφια ή δυνητικά υποψήφια. Σεβασμός επίσης των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων, στήριξη της κοινωνίας των πολιτών, στήριξη της, των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Τρεις βασικές σκέψεις εδώ πρόεδρε. Πρώτον, η συγγήτρια όπως και ο προηγούμενος συνάδελφος υπενθύμησαν την ανάγκη να διασφαλιστεί ένας αποτελεσματικός έλεγχος πολέμησης της διαφθοράς. Θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικά μέτρα ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει ένα σταδιακό πέρασμα στην άμεση διαχείριση των προενταξιακών μέσων από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην αποκεντρωμένη διαχείριση των χωρών οι οποίες ωφελούνται από αυτά. Είναι απαραίτητο λοιπόν να εισαχθεί και ένας μηχανισμός εξόδου από το μέσο αυτό δημιουργώντας μια μεταβατική περίοδο προς το Ταμείο Συνοχής και τα διαρθρωτικά ταμεία έτσι ώστε το μελλοντικό κράτος μέλος να προπαρασκευαστεί σωστά τη διαχείριση των μέσων. Έχουμε κάποιες εμπειρίες από ομάδες δράσης, task force, οι οποίες στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκαν στα διάφορα κράτη-μέλη και οι εμπειρίες αυτές μπορεί να είναι χρήσιμες. Είχε εφαρμοστεί και ένα πρόγραμμα στην Ελλάδα, το οποίο είχε προετοιμάσει τις, ε, τη δημοσιαδιοίκηση ε, στην είσοδό της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει επίσης να έρθουμε σε επαφή στενότερη με την κοινωνία των πολιτών, αποκαθιστώντας τις επαφές ανάμεσα στους πολίτες των διαφορετικών χωρών. Και πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα πιο σημαντικό ρόλο σε σχέση με το στρατηγικό κείμενο και αναφέρομαι εδώ στο 16, στο άρθρο 16, παράγραφος 18. Μου επιτρέπετε επίσης να εκφράσω μια προσωπική άποψη. Εγώ είμαι σκιώδης ε, σήμερα το απόγευμα στο θέμα, στο θέμα του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Θα ήθελα όμως να σας ζητήσω συγγνώμη ότι θα πάρω μέρος ψηφοφορίες, αλλά δυστυχώς αμέσως μετά θα πρέπει να αποχωρήσω και δεν θα μπορώ να είμαι παρόν. Ε, Euh, Ευχαριστώ Πρόεδρε, σύντομα, γιατί οι δύο αυτές εκθέσεις είναι συμπληρωματικές. Δημιουργούν ένα θέμα πάνω στο οποίο θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ προσεκτικά. Είναι το θέμα της συμπληρωματικότητας ανάμεσα στα ταμεία αυτά και στην πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης και ανάπτυξης της υπαίθρου όπως την ορίζει η Ευρωπαϊκή μας Ένωση στο εσωτερικό της Ένωσης. Αναγκαστικά βρισκόμαστε σε μια φάση επικάλυψης γιατί οι χώρες αυτές υποτίθεται ότι είναι προσανατολισμένες στο να ενταχθούν στην Ένωση. Συμφωνώ με αυτά τα οποία προτείνει η συγγήτρια. Την ευχαριστώ που εμένει στα θέματα της προστασίας των μειονοτήτων. Εγώ επιμένω ιδιαίτερο στην προστασία των εθνικών ταυτοτήτων μέσω και της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της επίσημης, δεν πρόκειται για κειμενόμενης γεωμετρίας βασικές αρχές, θα πρέπει να ισχύσουν και με τις χώρες γειτονίας και αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε όλες τις εκθέσεις. Πόσο μάλλον δε που στο προεντοξιακό μέσο υπάρχει δυνατότητα συγκεκριμένων μέσων και μέτρων Ξέρουμε τι γίνεται στα Βαλκάνια γύρω από αυτό, στις χώρες των Βαλκανίες στις χώρες της Βαλκανικές και θα θέλαμε κάπως πιο συγκεκριμένο τρόπο ε, και πιο συγκεκριμένες ενδείξεις για την οργάνωση των προγραμμάτων αυτών. Ευχαριστώ το λόγο έχει για την ανακεφαλαίωση η συγκεκριά μας η κυρία Γουκατσιεύσκα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις προτάσεις, τις συστάσεις, τις παρατηρήσεις. Συμφωνώ με περισσότερες από αυτές. Ε, το θέμα των υποδομών ή της πληροφορικής Νομίζω ότι αυτή είναι και η αχίλιος πτέρνα, όχι μόνο των υποψήφιων και δυνάμει υποψήφιων χωρών, είναι η αχίλιος πτέρνα ακόμη και των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορισμένων χωρών μελών, που προσπαθούν ε, συνεχώς ε, να βελτιώσουν την κατάσταση σε αυτά τα πεδία. Πάντως οι τροπολογίες μου λαμβάνουν υπόψη τις προτάσεις των σκιωδών εισηγητών, ιδιαίτερα για το θέμα της διαφθοράς ή της μεγαλύτερης δραστηριοποίησης ε, ε, των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις. Περιμένω τις τροπολογίες σας και ευελπιστώ ότι η τελική μορφή της γνωμοδότησης, η οριστική γνωμοδότηση θα τύχει γενικής υποστήριξης. Σας ευχαριστούμε κυρία Γουκασιεύσκα. Το μόνο που μένει να συμφωνήσουμε είναι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών και μετά τα σχόλια που κάνατε για την προηγούμενη, ας το κάνουμε λοιπόν και αυτό 3η Μαΐου. 3η Μαΐου στις 12 ακριβώς το μεσημέρι. Εδώ ας διακόψουμε την συνέδριαση του σημερινού πρωινού και επειδή έχουμε ψηφοφορίες το απόγευμα σας υπενθυμίζω να φέρετε τις ηλεκτρονικές σας κάρτες. Ευχαριστώ.